Dear Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα εργασίας ε, της Επιτροπής μας πριν από τις ε, διακοπές ε, τις οποίες τις αξίζουμε νομίζω, αλλά έχουμε ακόμα λίγη δουλειά Βλέπετε ότι είναι πολύ φιλόδοξη η ημερήσια διάταξη, οπότε θα σας παρακαλέσω για λίγη πειθαρχία. Και να υπενθυμίσω ότι έχουμε και μία ακρόαση και φροντίστε να είστε παρόντες. Δεν θέλω να είμαι μόνο εγώ εδώ με τους ειδικού μας. Περνάμε στο σημείο 1 για έγκριση της μερίσιας διάταξης. Υπάρχουν ε, κάποιες επιθυμίες για αλλαγές. Ε, όχι, οπότε εγκρίνεται. Δεν βλέπω κανένα να έχει κάποια αντίρρηση. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Ένα μήνυμα από τους διερμηνείς. Σήμερα είναι η 37η μέρα διαμαρτυρίας μας για την μονομερή επιβολή ε, συνθηκών εργασία από τη διοίκηση και δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να παραχωρήσουμε υπέρβαση ωραρίου σε αυτή τη συνεδρίαση. Σας ευχαριστούμε. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 3, ανακοινώσει τη ε, Προέδρου. Έχουμε σήμερα διερμηνία στα γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, τσεχικά, εστονικά, σλοβενικά, σλοβακικά, πολωνικά και ρουμανικά. Ως συνήθως η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο και περνάμε στις αποφάσεις των συντονιστών της 18ης Ιουνίου τις οποίες έχετε λάβει με email στις 20 του μηνός και εγκρίνονται αν δεν έχουμε κάποια αντίρρηση μέχρι τις 22 Ιουνίου. Μετά έχω να κάνω μία ανακοίνωση. Νομίζω ότι λάβατε όλοι σήμερα το πρωί ένα δωράκι, ένα βιβλίο συγκεκριμένα και σας είχα στείλει και ένα email με τις σχετικές πληροφορίες ε, για τον διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Βραβείου Λογοτεχνίας. Ε, έχουμε την δέκατη επέτειο και σκέφτηκαν οι διοργανωτές να κάνουν ένα διαγωνισμό μεταξύ των νικητών των 10 τελευταίων ετών και τους ζήτησαν να συντάξουν κάποια διηγήματα τα οποία θα κριθούν από μια κριτική επιτροπή και από εμάς τους βουλευτές. Οι υπεύθυνοι είναι σήμερα εδώ ε, στην Ευσό για να δώσουν ακριβώς αυτά τα διηγήματα τυπωμένα για να τα διαβάσετε στις διακοπές σας. Είναι στην πρωτότυπη γλώσσα και στα αγγλικά και όσον αφορά την ψηφοφορία υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες στο email που σας έχω στείλει και σας εύχομαι ήδη καλή διασκέδαση. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τους οργανωτές του Ευρωπαϊκού Βραβείου Λογοτεχνίας για τα βιβλία και καλή επιτυχία. Äh, ich finde, das ist ein Applaus Ναι. Χειροκροτήστε. Περνάμε λοιπόν τώρα στην ψηφοφορία. Έχουμε δύο προσωρινά αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου, ένα σχέδιο γνωμοδότησης και τις ε, τροπολογίες του προϋπολογισμού και δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε προτείνω να περάσουμε κατευθείαν στις ψηφοφορίες. Ξεκινάμε με το σημείο 4. Έχουμε τον συντονισμό κάποιων διατάξεων που αφορούν ε, νόμους ε, των κρατών μελών για την παροχή οπτικοακουστικών υπηρεσιών ποιος είναι υπέρ της οδηγίας αυτής από εμένα απλά ευχαριστίες ε, στους ε, συνεργασμούς μας και συγκεκριμένα στην Κατερίνα Φων και Χινοκούνα που έκαναν πάρα πολύ δουλειά, την Στεφανή Μπιατσόλη που είχε και γενέθλια χτες ε, και χρόνια της πολλά και βεβαίως σε όλους τους ε, συνεργάτες ε, των ομάδων, ε, των σκιωδών εισηγητών, αλλά και την γλωσσική υπηρεσία που μας βοηθάει στις διαπραγματεύσεις. Ήταν δύσκολες, αλλά νομίζω ότι καταφέραμε να φτάσουμε σε, κάποιες, σε κάποια καλά αποτελέσματα, σε κάποιους καλούς συμβιβασμούς για να εκπροσωπήσουμε και την θέση του Κοινοβουλίου στην οδηγία. Και πάλι λοιπόν ευχαριστώ για την επικοδομητική σας συνεργασία. Ζαμπίνε, θες να πεις κάτι? Βεβαίω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου ε, και, στην, και την κυρία Μπιαζόλη ε, και να πω πως ε, παρά τις δύσκολες συζητήσεις καταλήξαμε να επεξεργαστούμε έναν φάκελο ο οποίο ε, είναι θα έλεγα επικοδομητικός δεν είναι καθόλου απλό ο τριμερής διάλογο, ειδικά με την Εστονική Προεδρία η πρόοδος ήταν αργή θα έλεγα πιο επικοδομητική ήταν η συνεργασία με την Βουλγαρική Προεδρία οπότε θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερως και την Βουλγαρική Προεδρία που το έφερε εις πέρας στο εξαμεινό τη και χαίρομαι για το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ και τους ε, σκιώδεις εισηγητές που πράγματι ε, με περιέβαλαν με εμπιστοσύνη. Μάλιστα περνάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Geschlossen. Mit 19 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen. 19 υπέρ, 7 κατά, 2 αποχές εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υποθέτω ότι η τελική ψηφοφορία θα γίνει τον Οκτώβριο, πρώτη ή δεύτερη ολομέλεια, δεν ξέρω τώρα θα δείξει. Επόμενο αποτέλεσμα τριμερούς διαλόγου και αυτό δεν ήταν καθόλου απλό. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έχουμε την ψηφοφορία για την προσωρινή συμφωνία. Όπως είπα και αυτό δεν ήταν απλό. Χέλγα θέλεις τον λόγο. Ευχαριστώ. Πέτρα, να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους, τους ε, βοηθούς, ε, την δική μου βοηθό και τους υπόλοιπους. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, ειδικά όταν είχαμε τον τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο. Είχαμε μια πολύ καλά, καλή διαπραγματευτική ομάδα. Εμείς νομίζω τα πήγαμε καλύτερα από το Συμβούλιο και την ε, Κομισιόν, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάντα και χάρηκα ιδιαίτερο και νομίζω ότι ήμασταν πολύ επιτυχείς γιατί η πρώτη ανακοίνωση του Συμβουλίου ήταν μηδέν νέα λεφτά. Τώρα βεβαίως έχουμε 75 εκατομμύρια επιπλέον, βεβαίως θα θέλαμε ακόμη περισσότερα, αλλά καταφέραμε να εστιάσουμε στην μειονεκτική νεολαία και βεβαίως κυρίως να μιλάμε για εθελοντική εργασία, ελάχιστες ε, θέσεις ε, εργασίας πληρωμένες, ε, στις οποίες θα φελούσουμε να μην υπάρχει κατάχρηση και Πρόκειται για έναν αρκετά μεγάλο προπολογισμό στο επόμενο ΠΔΠ, το οποίο σημαίνει ότι τώρα οι νέοι μπορούν να πάνε σε ολόκληρη την Ευρώπη και παραπέρα για εθελοντική εργασία, να μάθουν κάποιες δεξιότητες, γλώσσες και κάποια άλλα πράγματα, κοινωνικές δεξιότητες και να επιδείξουν και κάποια αλληλεγγύη. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα πρέπει να ξεκινήσει γρήγορα το νέο πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ήταν πραγματικά εξαιρετική η διαπραγμάτευση που έγινε και νομίζω ότι για αυτό το φάκελο ήταν πραγματικά απαραίτητη. Ευχαριστώ λοιπόν. Νομίζω ότι φαίνονται τα καλά αποτελέσματα. Πάμε λοιπόν στην ε, ψηφοφορία. Και εδώ ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Geschlossen. Πέρας. Με 23 4 Με 23 ψήφους υπέρ, 4 ψήφους κατά και μία εποχή, εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στο σημείο 6, σχέδιο γνωμοδότησης για την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική της Ευρωζώνης. Εισηγητής ο κύριος Χουντής. Θέλετε το λόγο, κύριε Χουντή. Εντάξει. Άρα πάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία και ξεκινούμε με την τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Geschlossen. Πέρας. 16 με 12 απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική πρόταση 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό ήταν πολύ κοντά. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 14 προς 13 εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 27 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ γιατί δεν πολύ κατάλαβα. Geschlossen. Πέρας. 16 προς 11 εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. 28. Και αυτό σε δύο τμήματα. Υπέρ για το πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Και εδώ δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο. Υπέρ. Κατά αποχές να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοπαλία 13-13, απορρίπτεται. Τροπολογία 30, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31, υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 31. Πέρας ψηφορίας. 14-13 εγκρίνεται. 32 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ελέγχουμε. Πέρας 32-13. Απορρίπτεται με 14 ψήφους κατά και 12 υπέρ. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρο, προφορική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην τελική ψηφοφορία για το σύνολο της γνωμοδότησης, ονομαστική ψηφοφορία και άρχεται. Πέρας. 22 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά και 4 αποχές εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Σιγητή και ευχαριστώ τους σκιώδες. Πάμε στο σημείο 7. Σχέδιο προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Μοσονομικό του 2019 όλα τα σχέδια και έγκριση των τροπολογιών για το σχέδιο προπολογισμού. Πριν πέρασουμε στην ψηφοφορία, να ξεκαθαρίσω μια λεπτομέρεια. Στην περίπτωση των τροπολογιών του προπολογισμού δεν υπάρχει τελική ψηφοφορία, θα υπάρξει όμως στο τέλος μια ψηφοφορία ώστε να δώσουμε μια οριζόντια εντολή στον εισηγητή ώστε το σχέδιο προπολογισμού για όλες τις γραμμές που έχουν αλλάξει από το ε, Συμβούλιο να τις ε, αποκαταστήσει. Ο λόγος για αυτή την οριζόντια εντολή βρίσκεται στο ότι το Κοινοβούλιο στη διαδικασία την δημοσιονομική ε, κινείται προς τη θέση του Συμβουλίου. Αλλά τώρα θέλουμε να ψηφίσουμε πριν το Συμβούλιο ψηφίσει τη θέση του και γι' αυτό πρέπει να έχουμε εδώ την δυνατότητα να σχολιάσουμε και τις τροπολογίες του ε, Συμβουλίου. Γι' αυτό θέλουμε να δοθεί αυτή η οριζόντια εντολή στον εισηγητή μας. Ε, να δώσω το λόγο στον εισηγητή Μόρτεν Λόκεγκαρντ. Θέλει το λόγο, θέλει κάτι να πει. Παρακαλώ. Thanks, my colleagues, Mr. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τον κύριο Μόργανο, την κυρία Τρίπελ για την πολύ καλή συνεργασία. Ας προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ και σας Πρόεδρε και τους βοηθούς μου. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε στην ψηφοφορία. Υπάρχουν βόλικες τροπολογίες. Ξεκινούμε με την τροπολογία ε, συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην προφορική τροπολογία 1, η οποία βρίσκεται στην πέμπτη σελίδα, πάνω-πάνω. Προφορική τροπολογία 1, υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. 5769 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5770 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5778 υπέρ. 5778 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ωραία, να το ελέγξουμε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα δείτε ότι εγκρίνεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Geschlossen. Πέρας. 11 ψήφοι υπέρ, 6 κατά και 10 αποχές. Εγκρίνεται. Ε, 57-91 υπέρ κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. 57-92 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 57-97 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58-06 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58-07 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58-08 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην 57, 54 στην επόμενη σελίδα. 57-54 σελίδα 9 μέχρι επόμενη σελίδα. Υπέρ. Κατά αποχές πρέπει να το επαληθεύσουμε 57-54 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 13 υπέρ 13 κατά απορρίπτεται 57-68 υπέρ κατά αποχές δεκτή 57-79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5781 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5782 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5783 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5784 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57-87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Α, να το επαληθεύσουμε 57-87 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 57-88 υπέρ κατά αποχές δεκτή 57-98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57-99 υπέρ κατά αποχές δεκτή 58-13 υπέρ κατά αποχές δεκτή και 58-14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία για την οριζόντια εντολή για τον εισηγητή μας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 27 υπέρ, μία ψήφος κατά. Ο Μόρκεν Λόκεγκατ λοιπόν έχει οριζόντια έντολη. Καλή επιτυχία στις διαπραγματεύσεις εύχομαι. Σημείο 8. Νομοδότηση για τον Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019. Έχουν εγκριθεί όλα τα αιτήματα της Επιτροπής μας. Υπάρχει λοιπόν μία μόνο φάση παρά το ότι βεβαίως θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Η τελευταία φάση είναι η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για το συνολικό σχέδιο προϋπολογισμού του 2019 στο οποίο ουσιαστικά εξηγούμε τις τεχνικές τροπολογίες μας και στέλνουμε και πολιτικά μηνύματα στο Συμβούλιο. Πριν δώσω τον λόγο στον Μόρτεν Λόκεγκάρντ να σας πω πως η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι Παρασκευή 13 του μηνός στις 11 η ώρα και η ψηφοφορία είναι στις 3 Σεπτεμβρίου. Ελπίζω να μην σας τρομάζει η Παρασκευή και 13. Μόρτεν, έχεις τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως είπατε, η επόμενη φάση είναι η γνωμοδότηση για το προπολογισμό. Προφανώς θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις γραμμές του προπολογισμού που μόλις περάσαμε. Οπότε οι Σκιώδης και εγώ συμφωνήσαμε να υποβάλουμε τις τροπολογίες μας από κοινού με τις συμβαστικές προτάσεις. Αυτές οι τροπολογίες λοιπόν θα είναι για τα εξή σημεία και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος το βασικό πρόγραμμα που μας ενδιαφέρει, το Erasmus Συν, θα παραμείνει ε, με λιγότερα κονδύλια από ό,τι θα θέλαμε στο νέο προπολογισμό. Είναι πολύ χαμηλότερα από τις προσδοκίες του Κοινοβουλίου το Erasmus και στο επόμενο πουδουπού. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε αν θα το προκοδοτήσουμε παραπάνω στην επόμενη αναθεώρηση. Γι' αυτό ζητούμε αύξηση κατά 20% και σε τι τέσσερι δημοσιονομικέ γραμμέ του Εράσμου ΣΥΝ και για τι τωρινέ ανάγκε και για να αποστείλουμε ένα σαφέ πολιτικό μήνυμα για το πρόγραμμα στο μέλλον. Και αυτό είναι μια πολύ καλή ε, συμβαστική, πιστεύω, παρόλο που οι αριθμοί δεν είναι τόσο υψηλή όσο θα θέλαμε. Σημείο 2. Δημιουργική Ευρώπη, Creative Europe. Πρόγραμμα για την υποστήριξη της καλλιτεχνική δημιουργία στην Ευρώπη. Και αυτό δεν χρηματοδοτείται αρκετά και θέλουμε το επίπεδο να φτάσει στι φιλοδοξίε του προγράμματο. Σημειώνουμε ότι σε σχέση με το προ... υποπρόγραμμα για τα μέσα μαζική ενημέρωση πρέπει για να χρηματοδοτηθούν προγράμματα ποιότητα να έχουμε αύξηση κατά 44% τουλάχιστον. Για συμβαστικού σκοπού ζητούμε μια αύξηση 62% τουλάχιστον για να υπάρξει μεγαλύτερη στήριξη για το ευρωπαϊκό σινεμά ε, και τα σχετικά δίκτυα και να χρηματοδοτήσουμε τις προπαρασκευαστικές δράσεις χωρίς να διακινδυνεύσει χρηματοδότηση των ε, βασικών πραγμάτων. Τώρα, για το Ταμείο, το τομεακών προγραμμάτων και για το κεντρικό πρόγραμμα, ζητάμε 10% αύξηση για το πολιτιστικό υποπρόγραμμα επιπλέον 3, 3 ε, εκατομμύρια ευρώ ε, πάνω από το συνολικό κονδύλι για να ενισχυθεί η ατομική κινητικότητα και το σχετικό πρόγραμμα ε, των καλλιτεχνών και των δημιουργών στην Ευρώπη στο μελλοντικό πρόγραμμα. Τρία εκατομμύρια παραπάνω λοιπόν από τη συνολική αύξηση. Το επόμενο σημείο νέα διάταξη για την πολυθενία των μέσων μας και ενημέρωση και της ελευθεροτυπίας και ελευθερίας έκφρασης διατομεακά. Ε, Αυτό είναι απολύτως αναγκαίο βεβαίω, όμως για τη δημοσιονομική γραμμή η συνένεση στα οπτικοακουστικά και άλλα μέσα καθώς και τη δημιουργική βιομηχανία πρέπει να ενισχυθούν για να αντιμετωπίσουμε και τις ψευδείς ειδήσει με μια προσπάθεια αλφαβητισμού των μέσων και την άμεση στήριξη στις οργανώσεις που ε, ενισχύουν και παρακολουθούν την ελευθερία των μέσων και τον, ε, την πολυφωνία. Επίσης θέλουμε μια πλήρη αναθεώρηση όλων των δραστηριοτήτων στι γραμμέ του προπολογισμού για τα μέσα μαζική ενημέρωση, για να είμαστε βέβαιοι ότι επιδιώκουν του στόχου του και θα πρέπει να γίνει ε, τουλάχιστον στο επόμενο πίδι που, που, αυτό. Ε, για τι βασικέ δράσει και, ένα και ένα ποσό 4,2 εκατομμύρια επιπλέον από τι αναλήψει υποχρεώσεων για το 2019. Για την στήριξη του EuroNet και σε σχέση με όσα έχουν μείνει από το τρέχον που χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη λύση για το μελλοντικό τέτοιο πρόγραμμα. Για τη χρηματοδότηση από το 2020 και μετά έχουμε 8,4 εκατομμύρια χρηματοδότηση εδώ. Στο σημείο 4 πρέπει να ενισχύσουμε την αξία της Ευρώπης για τους πολίτες και να έχουν καλύτερη κατανόηση και αντίληψη της Ευρώπης και της ε, ιδιότητας του πολίτη. Θα πρέπει να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων πολιτών, λοιπόν. Λυπούμαστε που η νομοθετική πρόταση για τις νέε βεβαίω ε, διαδικασίε για την πρωτοβουλία των πολιτών δεν έχουν λάβει υπόψη τα αιτήματά τους. Το Κοινοβούλιο δεν είχε την ευκαιρία να παρέμβει στην ε, έγκριση της νέα πρότασης. Θέλουμε 10% αύξηση για τη διαδικασία αυτή βάσει του προγράμματο βάσει του νέου πολιτικού ε, δημοσιονομικού πλαισίου για να έχουμε τα απαραίτητα. Στο σημείο 5 για τις προπαρασκευαστικές δράσεις και τα πιλωτικά προγράμματα πρέπει να ε, χρηματοδοτήσουμε νέες καινοτόμες δράσεις. Πολλέ από τι προπαρασκευαστικέ δράσει και τα πιλωτικά προγράμματα που έχουν μεταδοτηθεί ω τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν αποδειχθεί επιτυχή για να ανοίξουν νέα καινοτόμα προγράμματα για την εκπαίδευση και την παιδεία. Γι' αυτό εκφράζουμε την δυσαρεσκιά μα για το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι σχετικέ διαδικασίε έγκριση δεν έδωσε χρόνο στο Κοινοβούλιο να τι επηρεάσει και να πει τη γνώμη του. Κάποιε φορέ τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποκειμενικά για να μην πω πολιτικά. Επηρεάζονται από τι θεσμικέ ε, προτιμήσει ε, και δεν είναι επαρκή. Θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη και στο μέλλον να το ξαναδούμε. Το έχω ζήσει τουλάχιστον δύο-τρει φορέ μέχρι τώρα. Να δούμε πώς ε, υλοποιείται αυτή η διαδικασία γιατί είναι επιφανειακή. Δεν ε, λειτουργεί καλά. Επιπλέον, και το λέω χωρίς να έχω συζητήσει με τους Κιώδης ακόμα, αλλά νομίζω θα συμφωνήσουμε, θα υποβάλω τροπολογία για να επαναλάβω την ανησυχία μας για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης χωρίς νομική, που ε, προβλέπεται χωρίς νομική βάση και αναμένοντα μια τελική απόφαση ε, για του πόρου που θα χρηματοδοτήσουν το σώμα. Παρομοίω, ε, με τι υπόλοιπε χρηματοδοτήσει για, την, ε, για τον προπολογισμό, θα προτείνω τροπολογίε για να ενισχυθούν οι συσχετισμοί τη χρηματοδότηση τη παιδεία και με άλλους πόρους ή δυνατόν από το ΕΦΣΙ, από το Horizon 2020 και 11 δις ευρώ είδαμε να μας λείπουν στο διάστημα 2007-2013, 2014-2020. Ε, προγράμματα ε, του με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Παρακαλώ ολοκληρώστε Μόργεν. Ναι, ναι, θα είμαι σύντομος για τα ευρωπαϊκά σχολεία επαναλαμβάνουμε την ανησυχία μας γιατί θέλουμε να ε, παρέχουν ε, ποιοτική διδασκαλία της αγγλικής ακόμη και μετά τον Brexit στα ανάλογα τμήματα ε, και να παραμένουν τα αγγλικά δεύτερη γλώσσα. Αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. So hearing Περιμένω τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να δώσουμε το λόγο στους χειόδες συγγητές. Δύο λεπτά το πολύ. Ο κύριο Στρογεύσκη πρώτα. Ε, κολέγα Λόκεγκάρτ, Συνάδελφε Λόκεγκάρτ, ευχαριστώ. Μας δώσατε μια πραγματικά ε, ενδελεχή εξήγηση των όσων πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα δεν είναι εύκολη η απόφαση που πρέπει να πάρουμε, αλλά οι βασικές προτεραιότητες για μας είναι το Erasmus Plus και εδώ έχουμε την αύξηση του 20%, 10% για το Creative Europe και για τον τομέα των ΜΜΕ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, το 22% είναι σημαντικό και 10% για την Ευρώπη των πολιτών. Θεωρούμε ότι χρειάζεται αλλαγή, αλλαγή συγγνώμη, στην προσέγγιση για αυτές τις γραμμές προπολογισμού και αξιοπιστία από την πλευρά της ε, Κομισιόν για την εφαρμογή όλων όσων έχουν συμφωνηθεί. Εδώ Έχουμε καταλήξει σε πολύ ευρύ συμβιβασμό για το θέμα αυτό. Δουλέψαμε πάρα πολύ καλά με τον εισηγητή. Και αυτό που ζητούμε είναι και αρκετά ε, ταπεινό. Είναι πολύ περιορισμένες οι ε, φιλοδοξίες που έχουμε. Θέλουμε απλώς μία αύξηση του προπολογισμού με βάση τις αναλογίες που έχουμε προτείνει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Λουίτζι Μοργάνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, του συναδέλφους και όδης εισηγητές για τη δουλειά μας ως τώρα. Πιστεύω η γνωμοδότηση που πρέπει να εκπονήσουμε θα επηρεαστεί και από τις τροπολογίες της Επιτροπής Προπολογισμών. Βεβαίω, ο εισηγητής Λόκεγκαρτ ήταν πολύ σαφής λέγοντα ποια είναι τα σημεία θετήρια για μα και ποια είναι τα σημεία που μπορούμε να υποχωρήσουμε. Θέλω να επαναλάβω ότι ω σοσιαλιστέ και δημοκράτε δεν είμαστε ικανοποιημένοι και δεν είμαστε ικανοποιημένοι ούτε ω Επιτροπή. Διότι ξέρω ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι ζητούσαν πολύ περισσότερα. Ο φόβο μα ε, σε κάποιο βαθμό ε, που έχει να κάνει με τη νέα ε, κατεύθυνση. Με συγχωρείς Λουίτζι, ε, πάλι το πρόβλημα. Μάλιστα, δεν είχαμε διερμηνία στα γαλλικά. Να επαναλάβω. Να ε, προσθέσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας, η δική μας μάλλον Επιτροπή Πολιτισμού, πάντοτε ομόφωνα ζητούσε περισσότερα κονδύλια σε σχέση με περικοπές που είχαν προαναγγελθεί από τη νέα Προεδρία του Συμβουλίου. Νομίζω στο νέο αυτό εξάμεινο το αυστριακό θα ληφθούν αυτέ οι αποφάσεις. Κάποιες ενδείξεις ακούσαμε και από πριν. Χθε είδαμε τι έγινε. Νομίζω ότι τα σημεία υποχώρηση ε, τα κατώτατα όρια που έχουμε προσπαθήσει με κόπο να κρατήσουμε σοσιαλιστές και δημοκράτες, έχουν να κάνουν με το ότι δεν θα μπορέσουμε σε καμία περίπτωση να εγκρίνουμε εάν δεν περάσουν. Και όπως είπε και ο συνάδελφος από το ΕΛΚ μόλις, Ε, επανειλημμένος μας τονίστηκε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ε, ε, ο τομέας του πολιτισμού θα λάμβανε μετά δεχματοδότηση χρηματοδότηση, τελικά θα είναι μια πάρα πολύ μικρή αύξηση. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορούμε να δεχτούμε τίποτα κάτω από αυτά τα όρια. Οτιδήποτε άλλο ούτε μπορούμε να το δεχτούμε, ούτε θα περάσει. Ευχαριστώ, Herr Ευχαριστώ. Ο μεγάλος καυγάς θα γίνει για το ΠΔΠ, γιατί αυτό θα δείξει τι μπορούμε να κάνουμε ετησίως με τον προπολογισμό. Οι σοσιαλιστές ψήφισαν υπέρ, εγώ ψήφισα κατά γιατί ξέραμε ότι θα μας δημιουργήσει προβλήματα με άλλα δημοσιονομικά προγράμματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι σε έναν ετήσιο προπολογισμό, και τώρα μιλούμε για τον ετήσιο προπολογισμό του 2019, πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι από τη μια, αλλά από την άλλη πρέπει να είμαστε και ρεαλιστέ. Γιατί βρίσκεται εντό ενό συγκεκριμένου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Αλλά τώρα πρέπει να πολεμήσουμε, γιατί πρέπει να το ενισχύσουμε. Δεν μπορούμε σε έναν ετήσιο ε, προπολογισμό να ζητάμε 100% αύξηση. Δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο αυτό από πολιτική οπτική. Οπότε εμείς σας ε, ε, ενθαρρύνουμε να προχωρήσετε. Ε, το 2019 λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε δυναμικοί, αλλά να ξέρουμε ότι ακριβώς ότι γνωρίζουμε και τι σημαίνει η αιτήσια διαδικασία. Οπότε εγώ συμφωνώ με την προσέγγιση του Μόρτεν, να είμαστε δηλαδή στην επίθεση, αλλά από την άλλη να δείξουμε ότι γνωρίζουμε και τι σημαίνει ισορροπία. Μιλήσατε για το Euronet Plus. Ε, νομίζω ότι είναι επίγον να πρικοδοτηθεί περισσότερο, γιατί συνδέεται και με τη συζήτηση που γίνεται για την ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα. Δεν το έχουμε σε όλα τα κρατη αλλά όταν υπάρχει τέτοιου είδου σύνδεση, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Και αυτό πρέπει να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και είναι σημαντικό και για τι εκλογέ του χρόνου. Πρέπει να φτάσουν ε, τα μηνύματα στου πολίτε μα. Και αυτό που είπε και ο, Μόργερ, ο Μόρτεν για, την, ε, για, τον, για τη διερευνητική δημοσιογραφία, για τι ψευδεί ειδήσει. Όλα αυτά πρέπει να τα παρακολουθούμε και πρέπει να ε, γίνει καλή δουλειά. Θέλουν να κάνουν καλή δουλειά και πρέπει να τους ενισχύσουμε. Και για το ε, ESC νομίζω ότι μπορώ να ακολουθήσω αυτό που προτείνεις. Θα ήμουν μάλιστα και πιο φιλόδοξη εγώ με το Συμβούλιο ειδικά, αλλά ξέρετε έχουν αυτούς τους πολιτικούς περιορισμούς στο Συμβούλιο. Ούτε ή άλλω αυτό είναι γενικό πρόβλημα και για το πολίτε δημοσιονομικό πλαίσιο. Οπότε α κάνουμε εμεί ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα τη ε, πολιτιστική διαφοροποίηση. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Μπίλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Σιγητέ. Σε ό,τι αφορά την αύξηση του προπολογισμού του Εράσμου ΣΥΝ για το 2019 και το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ωφελούνται πρώτα απ' όλα οι νέοι Ευρωπαίοι. Πράγματι, από το 2016-2017 το Εράσμου ΣΥΝ τίνει να ε, απασχολείται κυρίως με δράσεις ε, τις λεγόμενες ομάδες ε, του ευπαθούς πληθυσμού, ε, τις ομάδες του πληθυσμού, όπως τους Ισλαμιστές που πολλές φορές αποτελούν και κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα προβλήματα του προγράμματος, με πολύ ομιχλώδη όρους και, όρους και προϋποθέσεις. Και θα πρέπει, όπως είπε και ο εισηγητής, οι αθλητικές εκδηλώσεις να προαχθούν για να καταπολεμήσουμε την ξενοφοβία, τον ρατσισμό και την, να προάγουμε την καλή ένταξη. Όλα αυτά βέβαια δείχνουν τις καλές προθάσεις του εισηγητή, αλλά δεν είναι η βασική αποστολή του Ράσμου ΣΥΝ να προάγει την ε, εκπαίδευση και την απασχολησιμότητα των νέων. Θα πρέπει λοιπόν στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο ο τριπλασιασμός των δικαιούχων προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα προπολογισμό μόνο διπλάσιο να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Πρέπει να σκεφτούμε τις συνέπειες για τους νέους Ευρωπαίους οι οποίοι θα είναι πολύ λίγοι. Ε, πολύ λίγοι, αυτοί που θα μπορέσουν πραγματικά να ενισχυθούν στην κινητικότητά του. Και σε αυτό θέλω να προσθέσω ότι οι σχέσει συνεργασία, ιδίω με το Ευρωπαϊκό, οι διασυνδέσεις κυρίω με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, θα επιτείνουν αυτή την αρνητική τάση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας υπενθυμίσω ότι το Erasmus Plus δεν είναι πρόγραμμα απασχόλησης, είναι ρητά ένα πρόγραμμα κινητικότητας. Ε, ναι, αλλά η εκπαίδευση δημιουργεί θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα την Κομισιόν αν έχει να πει κάτι. Είναι εδώ. Ναι, ναι, παρακαλώ. Δύο λεπτά λοιπόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σιγητά, κύριε Σκιώδη. Κύριε Σκιώδη, Σιγητές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το σχέδιο προπολογισμού της 29 ε, Μαΐου για 166 εκατομμύρια, αύξηση σε σχέση με το 2018. Το σχέδιο αυτό προβλέφθηκε για να ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση των τρεχόντων προγραμμάτων καθώς και νέες πρωτοβουλίες με μεγάλη προσταθέμενη αξία, ευρωπαϊκή προσταθέμενη αξία, όπως ε, ευχήθηκε και ο πρόεδρος ο φιλόδοξος υπολογισμός της Επιτροπής σκοπό είχε να προάγει ακριβώς αυτούς τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την απασχόληση, την νεολαία, μαζί με την ε, διεύρυνση και την ασφάλεια και την άμυνα. Για την νεολαία, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την σταθερή σας στήριξη σε όσα έχουμε προβλέψει για τα τωρινά προγράμματα και για τις αυξήσεις που προτείνεται. Όπως ε, τονίζεται η επιτυχία των προγραμμάτων, Η επιτυχία των προγραμμάτων πολλές φορές δεν ε, ε, έχει αρκετά, η προσπάθεια για τους νέους δεν έχει αρκετά κονδύλια. είτε το πρόγραμμα της Δημιουργικής Ευρώπης, είτε τα προγράμματα για την απασχόληση δεν μπορούν να υποστηριχθούν αρκετά παρά τα καλά του ποσοστά επιτυχία, γιατί δεν υπάρχουν επιπλέον πόροι. Βεβαίω, πρόσθετα κονδύλια πάντοτε θα ήταν ε, επιθυμητά για να στηρίξουμε του δικαιούχου. Όπω προτείνεται, ο προπολογισμό του 2019 βασίζεται στα ποσά που προβλέπονταν στο Πουδουπού από το 2014-2020 κρίνονται ότι είναι μικρά τα ποσά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμω έπρεπε να κάνει δυσχερεί διαπραγματεύσει βάσει των διαθέσιμων ποσών και των περιθωρίων ανατίτλου του προπολογισμού. Αυτό δεν προδικάζει βεβαίω την δυνατότητα τη δημοσιονομική αρχή να ε, προτείνει αυξήσει εφόσον το επιθυμεί. Σα ευχαριστούμε για την πρόταση αύξηση Κάποιε κάποιες γραμμές των προγραμμάτων, όμω ήδη η αύξηση του 10% σε σχέση με το 2018 είναι πάνω από 60% σε σχέση με το 2014 στο κεφάλαιο 1. 2,1 ε, δις το 2019 σε σχέση με 2,3 και 1,5 το 2014. Το Erasmus Συν θα συνεχίσει στην πορεία του, άρα και θα μπορέσει να συνεχίσει τη δράση του που έχει μεγάλη ε, επιρροή. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ε, στα πλαίσια της δημιουργικής Ευρώπης, ο προπολογισμός που προτείνεται με άξιο 4% παραμένει στην γραμμή ε, των, ε, του πολιτισμού νομοσυνομικού πλαισίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόρτεν για να ολοκληρώσουμε. Έχετε τον λόγο. Θα είμαι, είμαι σύντομος, Πρόεδρε. Μια σύντομη παρατήρηση για όσα υπόθηκαν από Κιώδης και σας ευχαριστώ όλους. Νομίζω ήταν καλές οι συμβαστικές μας. Απλώς, σε σχέση με όσα είπε η κυρία Τρούπελ, η διαδικασία αυτή έφερε αντιμέτωπε δύο διαφορετικές σχολές στην ουσία. Κάποιοι θέλαμε μια πραγματιστική ρεαλιστική προσέγγιση και νομίζω ότι συμβαστική το απηχεί αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι επιτυχής και ευχαριστώ τους Κιώδης, συναδέλφους για αυτή την προσπάθεια. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα θέλαμε αύξηση στους αριθμούς, ότι δεν θέλουμε μεγαλύτερες φιλοδοξίες για αυτά τα προγράμματα. Νομίζω όλοι είμαστε εδώ φιλόδοξοι. Απλώς για οποιοδήποτε αμφιβάλλει, και εγώ προσωπικά τις έχω αυτές τις φιλοδοξίες, και θα φανεί αυτό και στις διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Να ε, χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις ε, ενωμένες μας δυνάμεις από την Επιτροπή αυτή, πηγαίνοντα στι διαπραγματεύσει για το πολιτέ. Διότι εκεί μπορεί κάτι να καταφέρουμε στου ε, αριθμού συνολικά. Να διατηρήσουμε λοιπόν την ενότητα τη Επιτροπή. Πάντοτε αυτή ήταν η δύναμή μα. Η ισχύ εν τη ενώση. Αυτό μας βοήθησε ως τώρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεργασία και ανυπομονώ για τις διαπραγματεύσεις. Äh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, 13 Ιουλίου, 11 η ώρα, η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες και ως εισηγήτρια για το σύνολο του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ σας διαβεβαιώ ότι θα είμαι πολύ φιλόδοξη εδώ και θα διαπραγματευτώ σκληρά με τους συναδέλφους, ε, αλλά νομίζω ότι συμφωνούμε με την βάση που εγκρίναμε τον Μάρτιο στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Δεν θα μας εγκαταλείψει βεβαίως ο προϋπολογισμός, ούτε του 19, ούτε το πι δελτα πι, οπότε θα μας απασχολήσει ξανά. Περνάμε στο σημείο 9. Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου. Έχουμε τον Κούρτσιο Μαλτέζε εδώ, ο οποίος ε, χτες δυστυχώς είχε κάποια προβλήματα με το αεροπλάνο. Όχι, δεν έχει δικό το αεροπλάνο. Όχι, όχι. Κάτι είχε συμβεί ε, με το, στο αεροπλάνο με το οποίο θα πέταγε. Οπότε υπήρχε κόλλημα Προθεσμία τροπολογιών είναι στις 12 Ιουλίου. Δεν βλέπω και κάποιον αντικαταστάτη του κυρίου Μαλτέζε, οπότε έχετε την έκθεση μπροστά σας και θα ήθελα να δώσω τον λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Τρεις είναι παρόντες αν βλέπω καλά. Ξεκινάμε τον κύριο Ντράγκητσι. Λοιπόν, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Αφού ζητούσαν χρόνια η ΜΚΟ μια σχετική νομοθεσία, η Κομισιόν παρουσίασε μια νομοθετική πρόταση που πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση. Χρειαζόμαστε μια σωστή προστασία των καταγγελόντων για να διασφαλίσουμε το δημόσιο συμφέρον ε, και να ενισχυθεί η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου, ειδικά στους ε, τομείς όπου μπορούμε να έχουμε παραβιάσεις οι οποίες βλάπτουν και το δημόσιο συμφέρον. Και ο δημόσιος και ιδιωτικός τομέας λοιπόν λαμβάνονται υπόψη και πραγματικές και οι δυνητικές παραβιάσεις ε, του νόμου καλύπτονται. Επίσης ε, ένα ευρύ φάσμα ατόμων ε, καλύπτεται και επίσης καλύπτονται και τυχόν αντίπινα Επινέες για αντίπινα προστασία και προστασία των κατηγορουμένων επίσης. Όμως αυτές οι πτυχές απαιτούν προσεκτική εξέταση και ενίσχυση της εμπιστευτικότητας επαρκή οικονομική και νομική βοήθεια και βεβαίως ε, να υπάρχουν και κάποιες εσωτερικές διαδικασίες, ένα ισχυρό πλαίσιο για τους καταγγέλλοντες. Αναμένω λοιπόν τον επικοδομητικό διάλογο και τη συνεργασία με τους άλλους εισηγητές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Evans. Ευχαριστώ. Δεν ε, έχω πάρα πολλά να πω. Μια πάρα πολύ καλή έκθεση. Πετυχαίνει την σωστή ισορροπία. Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αυτήν την οδηγία για να προστατεύσουμε τους ε, καταγγέλλοντες ε, ανθρώπους οι οποίοι ρισκάρουν την σταδιοδρομία τους για το δημόσιο συμφέρον. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε, να φροντίσουμε. Οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν αυτό το ρίσκο ε, για το δικό μας το συμφέρον να προστατεύονται και να έχουν μια σαφή απόψη για το τι μπορούν να κάνουν, τι ευθύνες έχουν και τις ευθύνες βεβαίως και των εργοδοτών για να προστατευτούν. Θα υποβάλω λοιπόν σχετικέ τροπολογίε, αλλά νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή έκθεση. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μπίλτ. Κυρία Μπίλτ, θέλετε να πείτε κάτι για την ε, οδηγία. Είστε εσκιώδη συζητήτρια. Συγχωρείτε. Πρόεδρε, ευχαριστώ οι καταγγέλλοντε μπορεί να προσφέρουν πραγματικά υπηρεσία καταγγελώντα παραβιάσει του δικαίου, αλλά και όλε τι ε, παράνομε και άτυπε δράσει όπω το κοινωνικό ντάμπινγκ. Πρέπει να προστατευτούν. Χρήζουν προστασία όχι μόνο σε επίπεδο σωματική ασφάλεια, αλλά και από νομική ε, σκοπιά. Διότι η οποιαδήποτε καταγγελία του μπορεί να ε, οδηγήσει σε εκφοβισμό τους και, ε, και μετά να μην επιτρέψει να αποκαλυφθούν και άλλα ε, κακό Υπάρχουν πολλά πρόσφατα διεθνή σκάνδαλα που έχουν λειτουργήσει σαν, ε, έχουν δείξει ότι λειτουργούν σαν ηλεκτροσόκ πολλέ φορέ οι καταγγελίε του. Γι' αυτό λοιπόν χρήζουν ουσιαστική προστασία. Όμω, όπω ο κ. Μαλτέζε ε, στο σχέδιό του λέει, δεν θα ήθελε να υπάρχει εφαρμογή ενό συγκεκριμένου προγράμματο, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βασιστεί στη γαλλική νομοθεσία που ζητά πρώτα να γίνει καταγγελία σε επίπεδο επιχείρηση, μετά σε επίπεδο δημόσια αρχή και τέλο το ίστατο επίπεδο να είναι εκτό εξαιρέσεων δημοσίω. Αυτή η πρόταση μου φαίνεται ε, σωστά εξορπημένη. Δεν θα πρέπει η προάσπιση των ε, καταγγελόντων να οδηγεί σε ε, ένα σύστημα συνολικής εμπλοκής θα πρέπει να προστατεύουμε τους καταγγέλλοντες ούτως ή άλλως χωρίς να περιμένουμε δημοσίως να φτάσουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της ίδιας της δικαιοσύνης και πρέπει να δούμε τι θεωρούμε ε, παραβίαση σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου ε, για να βεβαιωθούμε ότι οι καταγγέλλοντες ε, ε χρήζουν προστασίας δεν μπορούμε να περιμένουμε να αποφανθεί μια δικαστική αρχή πολύ αργά. Η σήμανση πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται καλή την πίστη, χωρίς τίποτε παραπάνω και ούτε να πάρουν ε, πολιτική διάσταση οι καταγγελίες των καταγγελόντων. Όταν η κοινή γνώμη θα έχει την άποψη ότι όλες αυτές οι καταγγελίες θα έχουν πολιτικές αποχρώσεις, δεν θα τους ακούει, οπότε η πρόταση αυτή δεν θα καταλήξει να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ίσα ίσα θα αποδυναμωθεί ο επιδιωκόμενος στόχος. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ, δύο λεπτά έχετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σημειώσαμε τα σχόλια της έκθεσης και τα όσα ακούσαμε σήμερα. Χαίρομαι που γενικώ το σχέδιο οδηγίας έτυχε υποστήριξης. Ένα σχόλιο σε σχέση με τη συμπερίληψη των αξιών της Ένωσης. Συμφωνούμε ότι ίσως αυτό μπορεί να διευρύνει υπέρμετρα το πεδίο εφαρμογής ε, και για σκοπούς νομικής ε, ασφάλειας θα ήταν δύσκολο να ορίσουμε πολύ ρητά και ξεκάθαρα αυτό το είδος των παραβιάσεων. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν είναι δοσίτης, άρα μπορούμε, δεν μπορούμε να το δώσουμε τον ε, λόγο. Να θυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι αύριο στις 12 και στις 24 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Πάμε τώρα στο σημείο 10. Συζήτηση με την Κομισιόν για την πολυγλωσία και την πολιτική επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλουμε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο, για το οποίο μας επέσαν την προσοχή οι Ευρωπαίοι πολίτες για τις πληροφορίες ε, των ε, ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θέλουν να τις βρουν στις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να τονίσω ότι η Επιτροπή μας ε, είναι καθήλυνα αρμόδια και επισήμω για το θέμα της πολυγλωσσίας και οι Ευρωπαίοι πολίτες νομίζω δικαίως ε, παραπονούνται ότι ψάχνουν αυτές τις πληροφορίες για τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες, για το πώς μπορούν να κάνουν την αίτησή τους, τι εργαλεία υπάρχουν για να τους βοηθήσουν, και θέλουν να τις βρουν στη γλώσσα τους, αλλά δεν είναι διαθέσιμες. Υπάρχουν 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο λίγες είναι αυτές τις οποίες μεταφράζονται στο σελίδες και προσφέρονται οι Ακόμα και τα πιο σημαντικά έγγραφα πολλές φορές υπάρχουν μόνο στα αγγλικά. Οπότε το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές αν τα κείμενα που τις αφορούν δεν υπάρχουν μεταφρασμένα σε όλες τις γλώσσες. Και ξέρουμε ότι το θέμα αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στην Επιτροπή μας. Και ως Επιτροπή σε έχουμε παραπονεθεί και έχουμε δείξει ότι αυτή η κατάσταση δεν μας ικανοποιεί. Γιατί σε, πολλές, αλλά σε πολλούς τομείς το θέμα δεν προχωράει. Έχει υπάρξει προσπάθεια να αλλάξει η κατάσταση, αλλά η, ε, Μιλούμε κυρίως για ε, προγράμματα που ασχολείται η Επιτροπή μας. Κοιτάξαμε και υπάρχουν ε, πάρα πολλά screenshots, αν θέλετε, να τα δείτε, από πολλές ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν μόνο στα αγγλικά οι τίτλοι μόνο έχουν ε, ε, μεταφραστεί και τα υπόλοιπα κείμενα που μπορεί να βρει κανείς είναι πάλι μόνο στα αγγλικά. Και αυτό ισχύει και για αιτήσει, για τα έγγραφα των ε, αιτήσεων και άλλα. Και παρόλο που Είμαστε επιτροπή που θέλουμε να φτάσουμε στα, στους πολίτες με τα προγράμματα αυτά, ε, ούτε εμείς δεν μπορούμε να τα βρούμε. Φανταστείτε οι άνθρωποι που δεν έχουν στη διάθεσή τους όλες τις υπηρεσίες μετάφρασης, να τους μεταφράσουν τα κείμενα, πόσο δύσκολο θα το βρίσκουν αυτό. Ειδικά για μεγάλα και δημοφιλή προγράμματα. Θα είναι πραγματικά καταστροφικό. Για το δικό μας τον τομέα δεν έχουμε λύσει επαρκώς το πρόβλημα και φυσικά ευχαρίστως θα ακούσουμε τους εκπροσώπους της Κομισιόν που είναι σήμερα εδώ και βεβαίως αν υπάρχει ενδιαφέρον και στους συναδέλφους μπορώ να στείλω όλα αυτά τα στοιχεία. Οι συνάδελφοι έκαναν πραγματικά πολύ προσπάθεια και ε, βρήκανε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα αρνητικά. Χαίρομαι λοιπόν που μπορούμε να έχουμε σήμερα μαζί μας τρεις εκπροσώπους από τρεις γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Κριστίνα Νάγκη πρώτα από την Γενική Διεύθυνση 5 Ο David Baker όχι δεν είναι εδώ, μισό λεπτό. Όλο αλλαγέ γίνονται. Λοιπόν, τη Βαλέρια Ντάρο έχουμε μαζί μας σήμερα από την Γενική Διεύθυνση TS1. Θα μπορέσετε ίσως να μας πείτε και τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά τα αρτικόλεξα. Η Φραντσέσκα Παγνοσίν που έχει να κάνει με την ε, συμπερίληψη των ε, ομάδων συμφερόντων από την ΕΑΚ και η Κριστίνα Νάγκη όπως είπα από την ε, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας που είναι υπεύθυνη για τις ευρωπαϊκές ιστοσελίδες. Πριν δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν, θα ήθελα καταρχάς να, δώσω, να θέσω εγώ δύο ερωτήματα, τα οποία θα μπορούσατε ίσως να συμπεριλάβετε στις απαντήσεις σας. Γιατί δεν έχουν μεταφραστεί αυτά τα σημαντικά έγγραφα για τους ε, Ευρωπαίους πολίτες και γιατί κρατάει τόσο πολύ μετάφραση αν γίνει και πώς μπορούμε επίσης να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει μετάφραση όλων αυτών χωρίς να υπάρχουν τόσο τραγικές καθυστερήσεις. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω το λόγο για 5 λεπτά στον καθένα και μετά θα κάνουμε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων. Δεν ξέρω ποιος θέλει να ξεκινήσει. Η κυρία Νάγκη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας και ευχαριστώ που μας δίνετε και την ευκαιρία να Σα παρουσιάσουμε το γλωσσικό καθεστώ των ε, ιστοσελίδων, αλλά και τις δυσκολίε που κι εμεί ε, οι ίδιοι αντιμετωπίζουμε, <laughs> ώστε να εξεύρουμε λύσεις για αυτή τη σημαντική πρόκληση. Είμαι εδώ με δύο συναδέλφους, τις παρουσιάσατε. Ε, μου ζητήσατε βεβαίως να σας ε, να πω τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά τα αρτικόλεξα. Η Βαλέρια είναι υπεύθυνη για τον, σχεδιασμό των μεταφράσεων στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης και η ε, Φραντσέσκα είναι υπεύθυνη για την ε, εκπαίδευση και τον πολιτισμό και Πώ ε, αυτές παρουσιάζονται στις ιστοσελίδε, όπως το είπατε και εσεί. Εγώ είμαι η ε, για τις ε, ευρωπαϊκές ιστοσελίδες. είμαι στη μονάδα επικοινωνίας της, ε, ευρωπαϊκής, ε, της Γενικής Διεύθυνσης. Και είμαστε και υπεύθυνοι για σχετικές επιμέρους ιστοσελίδες. Έχω, κάποιες, έχω μια παρουσίαση να σας κάνω την οποία θα την κάνω στα αγγλικά γιατί θα μου είναι και πιο εύκολο. Πολύ σύντομα λοιπόν. Να ξεκινήσω με κάποια αριθμητικά στοιχεία για αυτή την οικογένεια των ιστοσελίδων. Είναι σημαντικό να δείτε το μέγεθος και την περιπλοκότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά, αλλά και τα αποτελέσματα τελικά που επιτυγχάνουμε. Πέρσι είχαμε πάνω από 140 εκατομμύρια μεμονωμένους επισκέπτες που επισκέφθηκαν τις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με πάνω από 220 εκατομμύρια επισκέψεις. Αυτή η οικογένεια ιστοσελίδων είναι η δεύτερη στι στις ιστοσελίδες ε, κυβέρνησης και κοινωνίας ε, και είναι και η δεύτερη μεταξύ 3.700.000 σελίδων στο EU, στο domain.eu. Η παρουσία μας λοιπόν ε, στο διαδίκτυο είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προφανώς και για τους πολίτες. Ίσως αυτό να είναι το μόνο σημείο επαφής που έχουν με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Παίρνουμε λοιπόν τη δουλειά μας πολύ στα σοβαρά και θέλουμε να δώσουμε ε, τελευταίας τεχνολογίας ε, ε, πληροφορίες, υπηρεσίες για να μπορούν οι πολίτες να έχουν τις πληροφορίες που, έχουν στη διάθεση, που θέλουν στη διάθεσή τους. Έχουμε πολύ ξεκάθαρες κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες χρησιμοποιούν όλες οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες ετοιμάτων. Η μία είναι η μετάφραση περιεχομένου σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν το περιεχόμενο αυτό δεν μεταφράζεται προφανώς δυσκολεύει τη ζωή των πολιτών που θέλουν να προχωρήσουν την οποιαδήποτε υπόθεσή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίω έχουν ε, το δικαίωμα να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία των διαβουλεύσεων για την χάραξη τη πολιτική και επίση όταν είναι ε, νομικός απαραίτητο να γίνει οι μεταφράσεις. Και επίση όταν έχουμε σταθερό μόνιμο ε, περιεχόμενο στι ιστοσελίδε. Και έχουμε και άλλε περιπτώσει, βεβαίω, περιεχομένου όπου το περιεχόμενο αλλάζει ταχύτατα ή έχουμε πολύ συγκεκριμένο κοινό το οποίο αφορά το περιεχόμενο αυτό. Σε αυτές τις περιπτώσεις ενθαρρύνουμε τις υπηρεσίες να έχουν μια προσέγγιση με βάση συγκεκριμένα στοιχεία. Και εδώ θέλουμε να δούμε ποιο θα χρησιμοποιήσει τις ε, πληροφορίες και για ποιο λόγο. Ποιε γλώσσες ε, θέλουν, μπορεί να καταλάβουν καλύτερα οι χρήστες και επίσης ποια είναι η διαθεσιμότητα των πόρων για να μεταφραστούν και να, να μπορέσουν να διαχειριστούμε όλες αυτές τις ε, στο ιστοσελίδες και το πολύγλωσσο περιεχόμενο. Δείτε εδώ, ό,τι, είναι, ό,τι ε, άπτεται του νομικού περιεχομένου φροντίζουμε να είναι σε όλες τις γλώσσες και βάζουμε και τους συνδέσμους με το, με, στην υπηρεσία δημοσιεύσεων που έχει ούτως ή άλλως τις μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες. Ακόμα και αν η ιστοσελίδα δεν βρίσκεται, ε, δεν έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Οι σύνδεσμοι είναι πάντα μεταφρασμένοι. Για το νομικό τουλάχιστον περιεχόμενο. Επίσης, έχουμε δύο ιστοσελίδες πλήρως μεταφρασμένες σε όλες τις επίσημες γλώσσες, το Europa EU που είναι η διαθεσμική και η ιστοσελίδα της ε, Κομισιόν. Επίσης ε, έχουμε τις ε, μεταφράσεις σε όλες τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βεβαίως πάντα προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε. Έχουμε επενδύσει πολλά. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα για το τι πρόκειται να κάνουμε από εδώ και μπρος. Θα βελτιώσουμε την κάλυψη τη γλωσσική του, της ιστοσελίδας της ενημερωτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επόμενη επίσης εκδοχή του πόρταλ θα δώσουμε μεταφράσεις και σύντομες περιλήψεις ε, ώστε να ε, βελτιωθεί η ποιότητα των ε, διαθέσιμων πληροφοριών και επίσης προσπαθούμε να ενημερώσουμε και τις κατευθυντήρες γραμμές και να βοηθήσουμε διάφορες υπηρεσίες της Κομισιόν για, την, για να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, κυρίως για την προσέγγιση αυτή με βάση τα στοιχεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε κάνει μια μεγάλη έρευνα εδώ και κάποια χρόνια, η οποία αποτελεί τη βάση της δουλειάς μας για πολλούς τομείς Βεβαίως έχει να κάνει και με το γλωσσικό περιεχόμενο. Έχουμε πάνω από 100.000 απαντήσεις στην έρευνα αυτή, οπότε θεωρούμε ότι έχουμε μια πολύ στερεά βάση και αντιπροσωπευτική για τις ανάγκες των πολιτών από 211 χώρες. Αυτό λοιπόν που καταγράψαμε εδώ στο συγκεκριμένο πλαίσιο που συζητούμε σήμερα είναι ε, το ποιε είναι οι ενεργητικέ γλώσσε, οι πρώτε γλώσσε που χρησιμοποιούν οι πολίτε και οι δευτερογενεί, α πούμε, οι δεύτερη κατηγορία, ανάλογα με το γιατί θέλουν να ε, είναι σε επαφή με την ιστοσελίδα μα και να ψάξουν πληροφορίε. Το δεύτερο εργαλείο που χρησιμοποιούμε για αυτή την προσέγγιση με βάση της τα στοιχεία είναι τα ε, Web Analytics, όπου βλέπουμε τι ακριβώ γίνεται με το περιεχόμενο που ήδη είναι δημοσιευμένο στι ιστοσελίδε. Αυτό που μάθαμε τώρα από όλο αυτό το εγχείρημα είναι ότι ανάλογα με το πεδίο οι ανάγκε των πολιτών είναι πολύ διαφορετικές. Και βεβαίω σε τομεί όπω ε, η έρευνα ή τα χημικά, που είναι τεχνική, τεχνική τομή, α πούμε, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να καλύψουμε τις ανάγκες των πολιτών με αγγλικά. Αλλά αν είναι πιο προσωπικά τα θέματα, όπως ας πούμε συντάξεις, οικογένεια, η δυνατότητα εκεί των πολιτών να καταλάβουν ε, την, ε, τα αγγλικά είναι μάλλον μικρότερη. Εδώ ας πούμε βλέπετε την, ε, στη διαφάνεια τι γίνεται με το θέμα της, του πολιτισμού. τα αγγλικά ως ενεργητική αλλά και ως παθητική γλώσσα φτάνει περίπου το 90% των πολιτών. Αλλά βεβαίω ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει και ένα τεράστιο κενό. Το κενό αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό προσπαθούμε να δούμε πώ θα καλύψουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο το κενό αυτό. Οπότε έχουμε καταγράψει ποιε είναι οι γλώσσε που πρέπει να προσθεθούν για να μειωθεί το κενό αυτό. Εδώ βλέπετε ότι αν, αν, μειώσουμε, αν προσθέσουμε αγγλικά και, ε, γαλλικά και γερμανικά, συγγνώμη, μπορούμε να μειώσουμε το πεδίο, στο, το κενό αυτό στο 3%. Το 3% παραμένει σημαντικό, αλλά τουλάχιστον έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε την προσέγγιση αυτή. Τώρα, για τις γλώσσες που δεν είναι διαθέσιμες. εκεί περνούμε αμέσως στην αμέσως δια... επόμενη διαθέσιμη γλώσσα και αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ποιο είναι το ε, έγγραφο ή η ιστοσελίδα που δεν μπόρεσε να βρει στη γλώσσα του ο πολίτης που το έψαχνε. Εδώ ας πούμε βλέπουμε στην ε, ιστοσελίδα για, ε, για το μόνιμο περιεχόμενο ότι υπάρχει μια ιστοσελίδα η οποία δεν είναι μεταφρασμένη και για την και στην οποία δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον πολλοί πολίτε τη Ισπανία, για παράδειγμα. Οπότε κάνουμε συγκεκριμένη στοχευμένη μετάφραση πια, από εκεί και μετά, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει όντω μεγάλη ανάγκη. Ε, αντιμετωπίζουμε διάφορε προκλήσει, οι οποίε ε, σχετίζονται με του πόρου, με την ποιότητα του περιεχομένου. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε φυσικά όλου του διαθέσιμου πόρου που έχουμε και μιλήσατε και μόλις πριν για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οπότε η πτυχή, η οπτική του προπολογισμού είναι σημαντική. Πρέπει να δούμε το, την κάλυψη των γλωσσών σε σχέση με το κόστος της μετάφρασης και επίσης πρέπει να δούμε και την ποιότητα της μετάφρασης που είναι εξίσου σημαντικό τομέα. Η ε, βεβαίως ε, δεν είναι μόνο για τη μετάφραση που χρειαζόμαστε ε, τους πόρους, αλλά σε μια ψηφιακή εποχή που ζούμε πρέπει να επενδύσουμε ώστε να έχουμε τα σωστά εργαλεία. Κυρίως για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την αυτοματοποιημένη μετάφραση. Μόνο 20% προ το παρόν των ιστοσελίδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται στην ίδια πλατφόρμα, που σημαίνει ότι αυτό περιπλέκει ακόμη περισσότερο τα πράγματα και επίσης οι ψηφιακές επικοινωνίες σε σχέση με το πώς μπορούν να γίνουν λίγο πιο ομαδοποιημένες είναι άλλο ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λύσουμε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Φραντσέσκα. Ευχαριστώ. Χριστίνα, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Βλέπετε στην οθόνη την γλωσσική πολιτική για τα site ε, που έχει η γενική μας διεύθυνση, τρία που είναι σε όλες τις γλώσσες, τρία που είναι σε πέντε γλώσσες και δύο site που είναι διαθέσιμα στα αγγλικά. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα του Αθλητισμού, που αυτό περιέχει συνδέσμους ε, προς τις εθνικές σελίδες που είναι διαθέσιμες προφανώς στις εθνικές γλώσσες. Ακολουθούμε πλήρως την ε, γενική πολιτική της ε, Κομισιόν και λαμβάνουμε μέτρα για να υπάρξει ένας εξορθολογισμός ε, του περιεχομένου να προσπαθούμε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες στους χρήστες αλλά και να διευκολύνουμε τις υπηρεσίες μετάφρασης γιατί θέλουμε μια υπηρεσία που θα παρέχει καθολική υπηρεσία και να υπάρξει έτσι μια άρση των ε, εμποδίων στο γλωσσικό μέτωπο. Στο πλαίσιο αυτό αναφερθήκατε στην συμμετοχή στο πρόγραμμα και αυτό είναι η προτεραιότητά μας. Ε, θα ήθελα να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Ο οδηγός ε, του Εράσμους, ε, ξέρετε, πώς είναι, πώς να κάνει κάποιος αίτηση, δημοσιεύτηκε σε 23 γλώσσες την ίδια ημέρα σε ψηφιακή εκδοχή. Επιπλέον Έχουμε την συνεργασία με το εθνικό επίπεδο, με τις εθνικές υπηρεσίες, με το γραφείο της ε, Δημιουργικής Ευρώπης και σε αυτό το επίπεδο έχουν την υποχρέωση να δίνουν πληροφορίες στην εθνική γλώσσα αλλά και στήριξη στους πιθανούς χρήστες για να συμμετέχουν στα προγράμματα και αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον να παλύψουμε μια ανισότητα που οφείλεται στην χρήση κάποιας γλώσσας. Πιο Πιο πρόσφατα βελτιώσαμε κάποια από τα στοιχεία που δώσατε και εσείς, στις σελίδες του Erasmus, θα δείτε ότι κάποια τμήματα του ιστοτοπού έγιναν πιο λειτουργικά. Το μενού, το πώς να μπορέσει κανείς να σερφάρει στο site, οι σελίδες προσφέρονται σε όλες τις γλώσσες πλέον και επίσης μια σελίδα που είναι ε, πολύ σημαντική, πώς να θέσει κανείς να υποβάλει την υποψηφιότητά του για τους υποψηφίους που θέλουν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα δηλαδή. Βελτιώθηκε στο περιεχόμενό της και τώρα διατίθεται σε όλες τις γλώσσες. Εξηγείται σε όλες τις γλώσσες πώς μπορεί να γίνει η αίτηση και να συμμετάσχει κανείς. Για να ολοκληρώσουμε λοιπόν, για το site μας ακολουθούμε τη μεθοδολογία που μόλις ε, εξήγησε η Χριστίνα. Θέλουμε να υπάρχει αποτελεσματική χρήση των πόρων, διαρκής βελτίωση και έχοντας πάντοτε υπόψη τι υπηρεσίες θέλουμε να έχουν ε, στη θέση τους οι χρήστες του στο Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω πως έχετε λίγο στους ε, πόρους το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά είναι πραγματικά η κατάσταση αυτή ε, δεν είναι απολύτως ε, ικανοποιητική, αλλά τουλάχιστον τα βασικά των κεντρικών προγραμμάτων υπάρχουν σε όλες ε, τις γλώσσες. Δεν είναι και καμία φοβερή επιτυχία, αλλά όταν έχουμε ένα εγχειρίδιο για την Ευρωπαϊκή ημέρα αθλητισμού το να μεταφράζεται σε όλες τις γλώσσες εντάξει είναι κατανοητό αλλά όχι μόνο στην πρώτη σελίδα και μετά πατάμε τη δεύτερη σελίδα και υπάρχει μόνο στα αγγλικά γιατί βεβαίως θα, είτε δεν θα το πατήσει ο κόσμος ή βεβαίως αυτό οφείλεται στο ότι ε, τόσες ε, ε, και τόσες σελίδε υπάρχουν μόνο στα αγγλικά χωρίς να σημαίνει ότι γίνονται κατανοητές. Ε, έτσι είναι κάπως περίεργο αυτό. Έχουμε τώρα το μεγάλο πρόβλημα ότι πρέπει να τελειώσουμε ακριβώς 10.30 για να έρθει η Αυστριακή Προεδρία. Οπότε να δώσω τον λόγο στην Ζαμπίνε Φερχαΐν και την Σίλβια Κώστα. Παρακαλώ σύντομα και θα επανέλθουμε στο θέμα. Ζαμπίνε. Λοιπόν, για να είμαι σύντομη, αν δεν είναι ε, αγενές ε, κάτι τέτοιο κοιτάω τους αριθμούς σας, παραδείγματος χάρη λέτε τις προτινόμενες γλώσσες, ε, βλέπετε ότι τα γερμανικά είναι κάτω από το 10%, είναι μόνο κάτω από το 10%. Μα έχουμε 100 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη που μιλάνε γερμανικά ως μητρική στα 500 εκατομμύρια. Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Ε, ποιες είναι οι μητρικές γλώσσες, τι θα πει η προτιμόμενη γλώσσα. Πρέπει να κοιτάξετε τα νούμερά σας εδώ. Δεύτερον, το είπε η Πέτρα Καμερεβερτ. Μιλάτε για τελευταίες εξελίξεις ότι υπάρχουν ε, τα Εράσμους σε 24 ε, γλώσσες. Τέσσερα χρόνια από όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα, τέσσερα χρόνια από όταν προσπάθησε ο κόσμος ε, να λάβει μέρος στο πρόγραμμα και να κολλάει πάλι σε γλωσσικά εμπόδια, ειδικά από την Ανατολική Ευρώπη, ειδικά στις μικρές χώρες ειδικά σε αυτούς που θέλουμε ακριβώ να ε, αγγίξουμε, που δεν έχουν δηλαδή διεθνή εμπειρία. Ακριβώ είναι λυπηρό αυτό. Τέλος, ε, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού ή ο αθλητισμός μόνο στα αγγλικά, μόνο στα αγγλικά. αυτό είναι ε, πρόγραμμα για τους ε, μικρούς αθλητές, όχι για μεγάλους ε, μάνατζερ. Πώς θα γραφτούν αν υπάρχει μόνο στα αγγλικά και είναι και πολύ περίπλοκο. Δεν είναι μόνο οι πληροφορίες, αλλά απαιτούν και οι αιτήσει και οι απαντήσεις να δίνονται στα αγγλικά. Εντάξει, το βλέπουμε ότι ειδικά ακόμα και για επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με τα χημικά. Δεν μπορούν να λάβουν τις πληροφορίες. Η νομοθεσία ε, είναι μόνο στα αγγλικά και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να λάβουν τις πληροφορίες που θέλουν για πράγματα που αφορούν την ύπαρξή τους, την οικονομική έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει να εργαστεί περισσότερο η Κομισιόν στο γλωσσικό καθώς. Ε, Εκτός μικροφώνου. Ε, είναι εκτός μικροφώνου η ομιλήτρια. Ε, είναι διπλή η σημασία των προγραμμάτων αυτών. Δύο σχόλια και μια ερώτηση για την αυτοματοποίηση. Θα ήθελα να καταλάβω εάν η γλωσσική πολιτική και τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι κάτι που μπορεί να βελτιωθεί για να μπορέσει και η αυτοματοποίηση να είναι εύχρηστη. Εκεί που δεν χρειάζεται, συγκεκριμένη και ειδική μετάφραση για τα έντυπα, δεν κατάλαβα πολύ καλά. Είπατε για το Εράσμους ότι έχει ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Στον αθλητισμό ε, ε ακόμα πολλά πρέπει να γίνουν. Αλλά για τα θέματα πολιτισμού έχουμε καθυστερήσει σε σχέση και με το, την απόσταση, το κενό που είχαμε και για τι περισσότερε γλώσσε, το είπε και ο συνάδελφο Θα πρέπει λοιπόν να την καλύψουμε αυτή την απόσταση. Το θέμα είναι σε πόσο καιρό. Αυτό προσπαθεί να το δει και το Κοινοβούλιο. Και η ερώτηση είναι, είναι θέμα πόρων ή τεχνολογικών μέσων. Είναι πολλά τα site που έχουν μία ε, πλατφόρμα κοινή. Θα μπορούσαμε λοιπόν κάπως να επιταχύνουμε. και να ε, επιταχύνουμε λίγο την πρόσβαση στα προγράμματα σε όλες τις γλώσσες. Διότι αν είχαμε ένα τέτοιο στόχο κοινό, αν τον είχαμε εσείς και εμείς ως νομοθέτες, θα μπορούσαμε κάτι να πετύχουμε. Και τελευταίο, για τους εθνικούς φορείς. Η έκθεσή σας για τους εθνικούς φορείς, για να καταλαβαίνόμαστε. Ποιο είναι το κόστος μετάφρασης στις εθνικές γλώσσες επιβαρύνονται οι εθνικοί φορείς ε, το προπολογισμό αυτό ή ε, κάποια τμήματα μεταφράζονται, κάποια άλλα καθόλου. Τι συνεργασία υπάρχει. Πολλά από τα προγράμματά μας είναι σε συνεργασία με τους εθνικούς φορείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό για να ακούσουμε και απαντήσεις. Σας Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τις πληροφορίες αυτές. Και επειδή είμαι και εισηγητής ε, για το θέμα αυτό, θα ήθελα να πω ότι 60% των Ευρωπαίων δεν μιλάνε αγγλικά και στη χώρα μου, τη Βουλγαρία, φτάνει το 80% και πολλές ε, λαϊκιστικές ε, φωνές ακούγονται τα εκμεταλλεύονται αυτά. Εμείς μιλάμε τη γλώσσα μας ε, και τα λοιπά. Βλέποντας έτσι το θέμα, τι θα κάνετε για τον ρόλο των μικρών ε, γλωσσών. Και κάτι άλλο, στις 13 ε, Ιουνίου είχαμε μία συζήτηση για την αμοιβαία αναγνώριση των γλωσσικών ικανοτήτων τι σκόπευε να κάνει η Κομισιόν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρία λεπτά για τις απαντήσεις. Ε, θα επιμείνω σε αυτό. Όποιος θέλει. Να απαντήσω στην κυρία Κώστα για την αυτόματη μετάφραση. Η Επιτροπή εργάστηκε πολύ σε διάφορε υπηρεσίε τη Επιτροπή για να αναπτυχθεί ένα αυτόματο σύστημα μετάφρασης για όλες τις γλώσσες και με όλες τις δυνατέου ε, γλωσσικούς συνδυασμού, από και προς. Είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιείται πολύ και εσωτερικώ ε, στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης τη Επιτροπή ως βάση για να γίνει πιο γρήγορη η διαδικασία, να επιταχυνθεί η μετάφραση. Δεδομένη της ποιότητα όμω που θέλουμε να διατηρηθεί, όχι μόνο για την νομοθεσία, αλλά και για οτιδήποτε αποτελεί επικοινωνιακό υλικό για τους πολίτες και για τους ιστοτόπους, δεν μπορούμε να μην περάσουμε και από την μετάφραση με άνθρωπο. Η αυτόματη μετάφραση είναι ένα πρώτο κομμάτι, αλλά χρειάζεται και μεταφραστή. Δεν γίνεται ακόμα να το αφήσουμε. Και θα κοιτάξουμε το σύστημα αυτό να αναπτυχθεί περαιτέρω έχουμε προβλέψει διάφορες μηχανές που βασίζονται στο σύστημα των νευρώνων, τη μετάφραση των, ε, μέσω των νευρώνων με το σύστημα της τεχνητής ευθείας, κάτι που αναπτύσσεται ιδιαίτερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα και έχει απευθυνθεί και στις εθνικές αρχές, τους έχει γνωστοποιηθεί αν θέλουν να το χρησιμοποιήσουν. και προσφέρει και περαιτέρω ασφάλεια, περισσότερη ασφάλεια σε σχέση με άλλα συστήματα που κυκλοφορούν στην αγορά. Υπάρχει λοιπόν πρόοδο, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον ανθρώπινο παράγοντα για τη μετάφραση. Για τις ερωτήσεις για τις εθνικές αρχές. Οι εθνικές ε, αρχές και εθνικοί φορείς έχουν ε, υποχρέωση ε, να δημοσιεύουν στα site τους τα έντυπα, μεταξύ των οποίων αυτά για την υποψηφιότητα για το πρόγραμμα, ιδίως του Erasmus Στη σύμβασή τους υπάρχει ένας οδηγός για τους εθνικούς φορείς και προβλέπεται μια σειρά από κανόνες γι' αυτό. Έχουν επίσης την υποχρέωση οι εθνικοί φορείς, αν του ζητηθεί, να μεταφράσουν τμήματα συγκεκριμένα του υλικού. Για ό,τι αφορά τα έντυπα των προγραμμάτων, όλες οι υποψηφιότητε μπορούν να υποβληθούν σε όλες τις γλώσσες. Άρα δεν υπάρχει μπορεί να υπάρξει παθητική ανάγνωση και να συμβουλευτεί κανεί τα έγγραφα παθητικά, αλλά ενεργητικά μπορεί να υποβάλει την υποψηφιότητά όπω θέλει. Αυτό ίσχυε και για την ε, Creative Europe, για το πρόγραμμα που με ρωτήσατε. Νομίζω αυτά. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που σας πιέζω τόσο πολύ. Πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα. Ξέρετε, είμαστε ε, λίγο ανυπόμονοι εμείς εδώ και εξακολουθούμε να μην έχουμε ε, ικανοποιηθεί από τις απαντήσεις. Ξέρω ότι πολλά πράγματα υπάρχουν στα αγγλικά μόνο, αλλά ε, εγώ μπορώ να απαντήσω ας πούμε μόνο στα γερμανικά ή μόνο στα αγγλικά, στα ιταλικά. Αυτό σημαίνει ότι θα έχω καταλάβει καταρχάς στα αγγλικά τι σημαίνει η ερώτηση. Οπότε το δικό μας αίτημα είναι να φροντίσετε τα προγράμματα που όντως ε, είναι σημαντικά και για τα οποία δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι όλοι οι πολίτες που τα χρησιμοποιούν τα, τους ενδιαφέρον μίλαν αγγλικά. Ο συνάδελφος μίλησε για την κατάσταση στη Βουλγαρία. Και σε πολλα κρατημέλη κράτη-μέλη η κατάσταση είναι η ίδια. Ακριβώ λοιπόν για αυτά τα προβλήματα, για αυτά τα προγράμματα που θέλουμε να ασχοληθούν μαζί του οι πολίτε, να φροντίσετε να είναι μεταφρασμένα σε όλε τι γλώσσε. Γιατί εκεί θα, θα μπορέσουμε να επικεντρωθούμε. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να κάνετε κάποια πρόοδο. Ξέρω, ξέρω ότι προσπαθείτε να τα καταφέρετε. Σα ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Αλλά εμείς θα σας κάτσουμε στο σβέρκο, να είσαστε σίγουροι και σε κάθε βήμα θα παρακολουθούμε τι κάνετε ώστε να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Ευχαριστώ. So, wir können in unserer Λοιπόν, προχωράμε με την ημερήσια διάταξη και πάμε στο σημείο 11. Είναι μεγάλη μου χαρά που μπορώ σήμερα να καλωσορίσω την Αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου, η οποία μόλις ανελήφθη. έχουμε τέσσερις υπουργούς σήμερα το πρωί εδώ μαζί μας. οι οποίοι ασχολούνται με θέματα με τα οποία ασχολείται και η Επιτροπή μας. Και όλα αυτά βεβαίως είναι αρκετά διάσπαρτα στα διάφορα Υπουργεία, γι' αυτό και έχουμε σήμερα παρόντες τέσσερις ε, καθήλυν αρμόδιους υπουργούς. Οπότε, να ε, χαιρετήσω και να καλωσορίσω τον ε, Υπουργό Φάσμαν, που είναι Υπουργός Παιδείας και Επιστήμης, την Υπουργό Μπόγνερ Στράους, είναι υπεύθυνη για τα θέματα γυναικών νεότητας και νεολαίας και οικογένειας. Για το δεύτερο πάνελ θα ακούσουμε τον αντικαγκελάριο κύριο Στράχε, ο οποίος είναι υπεύθυνο για θέματα αθλητισμού και τον Υπουργό για την, τον κύριο Μπλούμελ, ο οποίος είναι Υπουργός στην Καγκελαρία για τα θέματα τα ευρωπαϊκά, την τέχνη και τα μέσα. Για κάθε υπουργό έχουμε αφιερώσει 10 λεπτά στο πρόγραμμά μας και μετά θα περάσουμε σε μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων. Θα συζητήσουμε λοιπόν. Αξιότιμε κυρία Υπουργέ Φάσμαν, αξιότιμη κυρία Υπουργέ Μπόγνερ Στράους, Καλώς ήρθατε. Είναι πραγματικά μεγάλη μας τιμή και χαρά μας να είστε εδώ. Είναι νομίζω το ότι η Αυστριακή Προεδρία αναλαμβάνει για, σε, σε μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και έχετε να αντιμετωπίσετε πολλές ε, προκλήσεις αλλά βεβαίως υπάρχουν και πολλές διεθνείς επίγουσες κρίσεις που πρέπει να διαχειριστείτε οι οποίες βεβαίως ε, θα καθορίσουν τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο. Εσείς λοιπόν έχετε αυτό το δύσκολο καθήκον, πρέπει να δείξετε πολιτικό όραμα και θάρρος για να αναλάβετε αυτές τις κοινέ προσπάθειες για τους τομείς της νεολαίας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, γιατί πραγματικά θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Είναι τομείς πολιτικής που νομίζω ότι ε, ε, ενδιαφέρουν πραγματικά τους πολίτες να υπάρξει πρόοδος. Ως πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής Πολιτισμού χαίρομαι πολύ που από κοινού μπορούμε να δουλέψουμε μαζί στους τομείς αυτούς. Νομίζω ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, συμφωνούν μαζί μου και φυσικά μπορείτε να βασίζετε στην απεριόριστη στήριξή μας. Ελπίζουμε ότι και εμείς θα μπορέσουμε να βασιστούμε στη δική σας ε, στήριξη για τα διάφορα θέματα που μας απασχολούν, κυρίως για την εκπαίδευση, την νεολαία, την, ε, ε, τον πολιτισμό κτλ. Κυρίως σε ό,τι αφορά την συζήτηση που θα γίνει στα, πλαίσια του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου, στα πλαίσια της συζήτησης για τον προπολογισμό. Ήδη υπάρχουν κάποια αιτήματα τα οποία ελπίζουμε, για τα οποία θα ελπίζουμε ότι θα δείξετε ευήκον ους. να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Φάσμαν για 10 λεπτά και μετά θα ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις και απαντήσεις και μετά θα ακούσουμε με τη σειρά την Υπουργό. Κύριε Φάσμαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές Ευχαριστώ και για την εισαγωγή. Πράγματι είπατε πολλά σωστά πράγματα και για την σημασία της ε, παιδείας ε, που είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουν οι εθνικές και η ευρωπαϊκή κοινωνία. Είναι κάτι το οποίο αφορά και το μυαλό και την καρδιά και βεβαίως ε, είναι κάτι το οποίο και προσωπικά με αγγίζει. Αν μου επιτρέπετε, στα 10 λεπτά μου θα αναφερθώ σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για εμάς και αυτό είναι οπωσδήποτε οι διαπραγματεύσεις για το Εράσμους. Το Εράσμους προτάθηκε ε, τον Μάιο από την Κομισιόν για το τι μορφή θα έχει από εδώ και μπρο ε, στο μέλλον και χαίρομαι για το ότι το πρόγραμμα εκμεταλλεύεται αυτήν την ε, ορμή που υπάρχει. Η εκπαίδευση ήταν ε, θέμα που μας απασχόλησε ήδη το 2017. Υπάρχει λοιπόν μια δυναμική την οποία πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Το Erasmus Plus είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα ε, προγράμματα, αν μου επιτρέπετε, το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα σύμβολο για την Ευρωπαϊκή Νεολαία η οποία μεγαλώνει μαζί ε, και επισκέφτεται άλλες πόλεις, ε, άλλα πανεπιστήμια. Είναι όμως συγκεκριμένα ένα μέσο για να προωθηθεί και μια ευρωπαϊκή ταυτότητα. Είχε ξεκινήσει πριν από 30 χρόνια και εκ 9.000 άνθρωποι έχουν λάβει μέρος. Και βεβαίως οι αξιολογήσεις δείχνουν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν έχουν χαμηλότερη ανεργία, υψηλότερες πιθανότητες να βρουν δουλειά, ψηλότερο εισόδημα και έχουν και μια κάποια ευρωπαϊκή συνείδηση. Οπότε είμαι αρκετά αισιόδοξο, αλλά και θέλω να προχωρήσει το Εράσμο. Σύμφωνα με την πρόταση θα ενισχυθεί, θα διευρυνθεί Νομίζω όλα αυτά είναι πολύ λογικά. Δεν υπάρχει κάποια επανάσταση αλλά μια μετεξέλιξη του προγράμματος ε, κάτι που είναι λογικό. Δεν υπάρχει και λόγος για μια εκβάθρον ανανέωση. Το πρόγραμμα είναι επιτυχημένο. Το πρόγραμμα θα έχει τρεις δράσεις κλειδιά. Η πρώτη είναι η κινητικότητα, η δεύτερη είναι η συνεργασία των Ιδρυμάτων και η τρίτη είναι η συνεργασία Υπουργείων, Κυβερνήσεων για την ανάπτυξη πολιτικών και ε, λοιπόν πρακτικών. Στην δεύτερη δράση υπάρχει και η αξιοσημείωτη ιδέα το, της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων να έχουν μια κοινή παρουσία και κοινά προγράμματα σπουδών, αλλά με έναν τρόπο πιο εντατικό από ό,τι συνέβαινε μέχρι στιγμής. Η ένωση αυτή, το European Universities όπως λέγεται, είναι αν θέλετε μια απάντηση στην δύναμη των παλαιών παραδοσιακών πανεπιστημίων και των πανεπιστημίων των ΙΠΑ. Θα ασχοληθούμε οπωσδήποτε με το θέμα αυτό και με την δράση αυτή, την πρόθεση της κινητικότητας για να μην ε, σπουδάζουμε μόνο, αλλά ε, να προωθηθεί ακριβώς ε, συνειδητά η κινητικότητα με τους μαθητές ε, και με όσους μαθαίνουν τέχνες, ε, ακριβώς ε, πρακτικές τέχνες, ακριβώς για να καταφέρουμε να εγγύξουμε και τα περισσότερα παιδιά για τις περισσότερες χρόνιες. Το πρόγραμμα Εράσμους λοιπόν είναι στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεών μας ελπίζουμε να υπάρχει μια θετική αντιμετώπιση των, θετικό των άλλων κρατών μελών και θα δούμε τώρα τι θα γίνει στις διαπραγματεύσεις. Δεύτερον, θα έχουμε το ζήτημα της αναγνώρισης, αναγνώρισης όχι μόνο στον ακαδημαϊκό τομέα όπου έχουμε ήδη πετύχει πολλά τα τελευταία χρόνια, έχουμε τη διαδικασία της Λισαβόνας και τον σχετικό κανονισμό. Κανονισμός, σύμβαση, σύμβαση, μάλιστα. Ορίστε. Και την Πολόνια, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Έχουμε προχωρήσει πολύ, αλλά βεβαίως ε, δεν έχουμε προχωρήσει πολύ στην αναγνώριση των ε, απολυτηρίων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ε, και αν θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης, θα πρέπει ακριβώς ε, να περιληφθεί και η δευτεροβάθμια ε, εκπαίδευση και όχι μόνο να περιοριστούμε στους φοιτητές και στους απόφοιτους πανεπιστημίων. Θα πρέπει τα χαρτιά να αναγνωρίζονται σε άλλη χώρα χωρίς εμπόδια και αυτό αφορά και την πρόσβαση μετά στη δεύτεροβάθμια εκπαίδευση και βεβαίως ε, να αναγνωρίζεται και όταν επανέρχεται κανείς στην δική του χώρα. Είναι μια πραγματική ε, κατάσταση και όποιος γνωρίζει την πραγματική κατάσταση θα συμφωνήσει ότι είναι ακόμα κάπως δύσκολα τα πράγματα. Τα πανεπιστήμια λένε ε, δεν ξέρω αν αυτό το οποίο μάθατε εκεί είναι τόσο καλό με, σε σύγκριση με αυτό το οποίο διδάσκουμε εμείς εδώ και επίσης δεν ξέρω αν ε, αυτοί οι οποίοι αποφυτούν από το Λύκειο εκεί είναι εξίσου ικανοί με τους δικούς μας ε, εδώ. Ε, αντιλαμβάνομαι αυτήν την επιφυλακτικότητα, την γνωρίζω καλά και χρειάζεται νομίζω ένα πιο δεσμευτικό μέσο για την αμοιβαία αναγνώριση. Υπάρχουν καλά παραδείγματα τέτοιων αυτόματων αναγνωρίσεων. Οι χώρες Benelux έχουν προηγηθεί, οι σκανδιναβικές χώρες, οι βαλτικές χώρες μεταξύ τους. Πρέπει να ακολουθήσουμε λοιπόν αυτά τα υποδείγματα. Οπωσδήποτε θα έχουμε επιτυχίες που θα αφορούν την διασφάλιση της ποιότητας ε, και υπηρεσίες ε, σχετικές και βεβαίως θα έχουμε και κάποια άλλα σημεία στα οποία θα δώσουμε βάρος ε, διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών είναι κάτι το οποίο επίσης θα μας απασχολήσει. Έχουμε επίσης το θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης, ε, στρατηγικές εφαρμογής, ε, ψηφιακή εκπαίδευση, μεταρρυθμίσεις εκπαιδευτικές, πάντα με τον σκοπό να έχουμε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης. Βλέπετε ότι έχουμε ε, ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ελπίζω να συνεχίσουμε τις ε, συζητήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι μας ε, χαροποιεί το ότι έχετε ως πρώτη προτεραιότητα το Εράσμους αλλά και τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρατε. Θα ξεκινήσω τώρα με τις ερωτήσεις. Ζαμπίνε Φερχάιεν. Αναφέρατε το πρόγραμμα Εράσμου, το οποίο θα ενισχυθεί από την Κομισιόν. Ε, γνωρίζετε κύριε Υπουργέ ότι αυτή η ενίσχυση ουσιαστικά αποτελεί την ε, επιβεβαίωση των δύο ή τριών προηγούμενων ετών και, σημαίνει, και δεν σημαίνει τελικά όντως μεγαλύτερη ενίσχυση σε σχέση με αυτό που ζητάμε εμείς. Έχουμε ξεκινήσει αυτή την περίοδο προπολογισμού, έχουμε ολοκληρώσει, έχουμε ε, φτάσει σε ένα σημείο της χρηματοδότησης, αλλά δεν ε, αποτελεί βελτίωση του ε, status quo. Γιατί μιλούμε για ένα ανώτατο όριο 20% των επιλέξιμων αιτήσεων για το πρόγραμμα Εράσμους. Αυτό δεν σημαίνει και τεράστια βελτίωση. Γιατί και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε αιτήσει πολλέ οι οποίε θα πρέπει δυστυχώ να απορρευθούν. Αυτό σημαίνει ότι στην δομή του προγράμματο Εράσμου θα πρέπει να μπει και το πρόγραμμα για, το, για τα εισιτήρια Interrail. Οπότε σας ρωτώ, είσαστε έτοιμοι να ξεκινήσετε με κάτι τέτοιο, ώστε δηλαδή ο προπολογισμό για το Εράσμος όχι απλώ να διπλασιαστεί αλλά να ε, αυξηθεί σημαντικά. Γιατί σωστά είπατε ότι είναι το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα, αλλά θέλουμε να παραμείνει επιτυχία στο πρόγραμμα του Εράσμού. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να δημιουργούμε άλλα προβλήματα στους ε, ετούντες. Επίσης, η ενίσχυση των δραστηριοτήτων και στην επαγγελματική εκπαίδευση για τα προγράμματα ΒΕΤ. Ενίσχυση τέλο πάντων του παλιού Κομένιου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Είναι, υπήρχε το Λεωνάρντο, το Κομένιου, μετά τα συγχωνεύσαμε τα δύο και υπήρξε αυτή η ε, χρηματοδότηση, αλλά πάντα σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με την ε, ε, ανταλλαγή των πανεπιστημιακών φοιτητών. Εμείς θεωρούμε ότι και στον τομέα αυτό θα πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα, όχι μόνο για τους αποφύτους των πανεπιστημίων, αλλά και για, τον, για την επαγγελματική κατάρτιση και εκεί θα πρέπει να ενισχυθεί αυτό ήδη από τα χρόνια της παραδοσιακής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υπάρχει ε, άρνηση για την ε, αύξηση του προπολογισμού για το επόμενο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά πρέπει να υπάρξει άμεση ε, αύξηση ακριβώς για το πρόγραμμα αυτό. Γιατί εκεί χρειάζονται τα περισσότερα κονδύλια. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Αμέσως, αμέσως. Θα κάνουμε πινκ-πονγκ. Σε, κυρία Ευρωβουλευτά, συμφωνώ με τα όσα είπατε για το Erasmus, το είπα και εγώ στην εισαγωγή μου. Αυτό το 20% δεν το καταλαβαίνω, δεν κατάλαβα ακριβώς πώς το εννοήσατε. Εγώ ήμουνα αντιπρίτανης σε ένα μικρό πανεπιστήμιο στη Βιέννη για έξι χρόνια και παρακολουθούσα τα προγράμματα τα διεθνή. Ποτέ δεν χρειάστηκε να απορρίψουμε κάποιον φοιτητή. Σχόλια χωρίς μικρόφωνο. Ναι, αλλά το 100% πού είναι. Μιλάτε για έγκριση 20% εσείς. Ε, πρέπει να μου το εξηγήσετε νομίζω. Και επίσης πρέπει να μου εξηγήσετε και κάτι άλλο. Γιατί αυτή η ονομαστική αύξηση των 15 δισεκατομμυρίων που είναι 30 δεν, έγινε, δεν είναι σημαντική αύξηση. Ε, δεν καταλαβαίνω. Λογιστικά είναι σημαντικό το ποσό είναι σημαντική αύξηση. Θα μπορούσε κανεί να πει ότι μπορεί να πάει και παραπάνω. Αυτό να το καταλάβω. Δεν έχω εγώ να πω τίποτα ως προς αυτό, δεν έχω καμία αντίρρηση να υπάρξει και άλλη αύξηση. Αλλά οι διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει, ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να τις προκαταλάβουμε, ούτε χρειάζεται. Επίσης, χρειαζόμαστε αύξηση των, ε, ε, ε, φοιτητών που βρίσκονται στα επαγγελματικά προγράμματα. Και για την κινητικότητα των φοιτητών, νομίζω ότι υπάρχει και ένα επίπεδο το οποίο ένα οριακό ας πούμε επίπεδο αλλά ακόμα δεν είμαστε εκεί έτσι όπως ε, δομούνται οι εγκύκλοι και όπου μπορεί να υπάρχει ένα παράθυρο κινητικότητας, είναι καλό, έτσι ώστε να μην οδηγεί η κινητικότητα σε καθυστέρηση των σπουδών, αλλά σε εμπλουτισμό αυτών. Ούτως ή άλλως ε, υπάρχουν ε, θέματα οργανωτικά ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα για το, για το Εράσμους. Ευχαριστώ. Ε, ναι, μιλούμε για, τα, για τις αιτήσει, κυρίως Μιλούμε για το παλιό πρόγραμμα κομμένιους με τις ε, εταιρικέ σχέσεις μεταξύ σχολείων, αλλά μιλούμε και για τον τομέα της νεολαίας και αυτή την πτυχή του Εράσμους που αφορά στη νεολαία, όπου πάντα project απορρίπτονται και όταν λέμε ότι δεν αρκεί αυτή, αυτός ο διπλασιασμός, θα πρέπει να δούμε αν το 2020, που είναι το τελευταίο προγραμματικό έτος, και έχουμε και το backloading το οποίο ούτως ή άλλως αυξάνεται. Αν λοιπόν στο τελευταίο, αν βάλουμε το τελευταίο έτος ως το 2020 και το ξεπεράσουμε, τότε νομίζω ότι θα βρεθούμε στα 24 δισεκατομμύρια. Έρχονται άλλα 16 τα οποία επίσης πρέπει να τα συνυπολογίσουμε. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ναι είναι αύξηση μεν, αλλά δεν είναι η αύξηση που τελικά χρειαζόμαστε για να μπορεί το πρόγραμμα αυτό να γίνει ακόμη πιο επιτυχές. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Σίλβια Κώστα, δύο λεπτά το πολύ. Κύριε Υπουργέ, από την πείρα σας ως, ε, ως αντιπρίτανη, με ακούτε, ωραία, ωραία γιατί τα λέω Ιταλικά, έλεγα από την πείρα σα ω αναπληρωτή ε, πρίτανη, ε, Μπορείτε να μα πείτε πολλά ενδιαφέροντα, γιατί φαντάζεστε πόσο προσφυλή μα είναι αυτό το τόσο ουσιαστικό για την Ευρώπη. Δεν επενδύουμε στην εκπαίδευση και την παιδεία των νέων και νέων και στα εκπαιδευτικά συστήματα. Ε, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα χάσουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Ο πολιτισμό, η παιδεία, η εκπαίδευση, η έρευνα και η οικοδομία είναι η καρδιά της Ευρώπης, είναι η βασική δουλειά της Ευρώπης. Εμείς και το συμπεριλάβατε στις προτεραιότητά σας βλέπω, που είναι και πολύ συγκεκριμένε και επί της ουσίας. Βλέπουμε να αλλάζει ο ρυθμός στις εκπαιδευτικές πολιτικές στην Ευρώπη να αλλάζει το κλίμα. Και ελπίζω η Αυστριακή Προεδρία να το αναλάβει αυτό το κλίμα και να το ε, παρακολουθήσει στενά ε, υπάρχει ε, διάθεση για έναν ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευση. Όχι μόνο για την ανώτερη εκπαίδευση, αλλά γενικότερα για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Στις συστάσεις που αναφερθήκατε, ελπίζουμε να περιληφθεί αυτό στι προτεραιότητε τη Προεδρία σα και να δώσετε όθηση στι προσπάθειε για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων και ίσως για τη δημιουργία ενός οργανισμού. Θα ήταν ε, ενδιαφέρουσα αυτή η ιδέα για να υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε σχέση με το πρόγραμμα. Σε αυτό το πρόγραμμα που έχετε την Προεδρία θα γίνουν οι πρώτες σημαντικές διαπραγματεύσεις για τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Για μας είναι σαφές ότι το Εράσμους είναι μια μαγική κουβέντα που καλύπτει όμως πολλές διαφορετικές προεκτάσεις, οι οποίες κάπως πρέπει να επανασταθμιστούν για τις επαγγελματικέ δεξιότητες, για τις πολιτικές της νεολαίας που καλύπτει το Εράσμους, για την δυνατότητα πρόσβασης συνολικά και θα ολοκληρώσω γρήγορα. Θα πρέπει να εκριθεί και πάλι το Εράσμους Μούντους. Ελπίζουμε να έχουμε την Αυστρική Προεδρία στο πλευρό μας αυτό. Και θα πρέπει να διευκολυνθεί η δυνατότητα για νέα παιδιά που δεν έχουν ε, χρηματικά μέσα να έχουν πρόσβαση. Θέλουμε να στηρίξουμε τους Ευρωπαίους φοιτητές και να δοθεί έμφαση και στις εταιρικές σχέσεις μεταξύ σχολών, ενώσεων, επαγγελματικών ενώσεων και των ε, λεγόμενων key action των εταιρικών σχέσεων το Εράσμος για μας πρέπει να τριπλασιάσει τα χρηματοδοτικά του μέσα. Αυτό έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο κατά ευρεία πλειοψηφία. Ελπίζουμε να γίνει δεκτό το έτοιμά μας. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ κύριε Κώστα για τις ερωτήσεις. Ελπίζω να έχω καταλάβει όλα όσα είπατε. Καταρχάς για το Εράσμους απλούστευση του Εράσμους, ανεξάρτητα από την οικονομική προκοδότηση, έτσι ώστε να γίνει πιο προσβάσιμο για τους φοιτητέ, για τους νέους, για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Δεν διαφωνώ καθόλου. Είμαι απόλυτα σύμφωνος μαζί μας. Το, αν δούμε και τις συμφωνίες μάθησης, το Εράσμος ούτως ή είναι ε, περίπλοκο. Χρειάζεται να γίνει μια συμφωνία μάθησης πριν πάω εγώ στην άλλη χώρα για να σπουδάσω αν ε, λήξει αυτή η συμφωνία ε, πρέπει να ξανακάνω νέα συμφωνία, πρέπει το ε, εκπαιδευτικό ίδρυμα της άλλης χώρας να έρθει σε συνεννόηση με το εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας μου, είναι πολύ περίπλοκο όλα αυτά. Όντω υπάρχει η φιλοδοξία να είναι επιτυχία το Εράσμος, το είπα και θα το ξαναπώ, γιατί είσαστε ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γυρνάτε πίσω στις χώρες σας Οπότε πείτε στα πανεπιστήμια σας ότι πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις για, τις, ε, για να μπορέσει να λειτουργήσει, να λειτουργήσει το Εράσμος. Αυτές οι προϋποθέσεις ε, για τις, ε, μέσω των εγκυκλίων είναι πάρα πολύ σημαντικές για το, και μάλιστα πολύ πιο σημαντικές από το αν θα πάρει ο φοιτητή 400, 450, 500 ευρώ για το Εράσμος. Γιατί ξέρουμε ότι οι εγκύκλοι όταν είναι τόσο αυστηρές δεν επιτρέπουν θέσεις για το Εράσμος. Δεύτερο ερώτημα. Είναι το θέμα της αναγνώρισης. Αναγνώριση ως προϋπόθεση για, την, ε, για τον κοινό ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό χώρο. Νομίζω ότι όλοι εδώ στην αίθουσα συμφωνούμε ως προς αυτό. Η υπηρεσία τώρα νομίζω είναι λανθασμένη έκφραση ε, ή τέλο πάντων εγώ δεν το καταλαβαίνω έτσι. Δεν πρόκειται να φτιάξουμε νέα υπηρεσία ή οργανισμό. Απλώς χρειάζεται μια διαδικασία αναγνώρισης η οποία θα λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί και η αντίστοιχη για τα πανεπιστήμια. Αυτό χρειαζόμαστε και για τα διπλώματα των γυμνασίων τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό. Χρειάζεται εμπιστοσύνη των κρατών μεταξύ τους έτσι ώστε τα ε, ε, ε πτυχία των, ε, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να είναι ποιοτικά. Χρειαζόμαστε φιλοδοξία από τα κρατημέλη, ώστε η, δευτερο, η δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους να μπορεί να εξασφαλίσει μια ποιότητα και αν τα έχουμε καταφέρει και τα δύο, και τη διαφάνεια και την ποιότητα, στον τομέα αυτό της, των ε, διπλωμάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τότε πιστεύω ότι κάτι θα έχουμε κερδίσει. Θα μπορέσουμε ίσως να απαντήσουμε στο θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης ή τέλος πάντων θα μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε. Και μετά μιλήστε για ένα τρίτο θέμα, για το Erasmus Mundus. το Erasmus Mundus θα συνεχίσει να υπάρχει και είναι κάτι το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μένα προσωπικά. Το Erasmus δεν θα πρέπει να γίνει απλώς πιο συμπεριληπτικό, θα πρέπει να γίνει και πιο διεθνές. Γιατί ανήκει κυρίως στην ευρωπαϊκή, ε, στα ευρωπαϊκά σύνορα. Και εκεί σταματά. Το Erasmus Mundus ανοίγει την πόρτα στον κόσμο σε τρίτες χώρες. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πραγματικά σημαντική η φιλοδοξία. Και ελπίζω βεβαίως ότι θα συνεχίσει να υπάρχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει τώρα η εξή δυσκολία. Εφτά συνάδελφοι έχουν ζητήσει τον λόγο. Έχουμε όμως ελάχιστο χρόνο. Σας παρακαλώ λοιπόν να σκεφτείτε πως ε, θα μπορούσατε να απευθύνετε κάποια ερωτήματα προς την κυρία Μπόργνερ Στράους και έχουμε και άλλους υπουργούς. Θα δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε. Χέλγα Τρίπελ λοιπόν. Θα είμαι σύντομη λοιπόν. Θα εστιάσω σε μία συγκεκριμένη ερώτηση, αν και έχω κι άλλες. Ο προπολογισμός και το πει. Το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο Μιλήσατε για την ποιότητα και την ε, συνεργασία. Ναι, σωστό. Αλλά βεβαίω θα πρέπει η αστιακή κυβέρνηση ως Προεδρία να δει το θέμα του ύψους του ΠΔΠ συγκεκριμένα για την εκπαίδευση. Η Ζαμπίνε έχει δίκιο όταν λέει ότι το backloading. Αυτό δεν θα κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει και απαιτείται για τους νέους. Ε, πρέπει όμως να γίνει αυτό εάν θέλουμε πραγματικά να ασχοληθούμε με το μέλλον των νέων στην Ευρώπη. Ξέρουμε το τι γίνεται ειδικά στην Ήπεθρο και πώς καταλήγει αυτό πολιτικά. Εντάξει, μπορεί να σας ικανοποιεί εσάς περισσότερο από ότι εμένα, αλλά ψηφιακά δεν έχουν πολλές ευκαιρίες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουν όσο το δυνατόν καλύτερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία το Erasmus Plus. Γι' αυτό θα πρέπει να αντιληφθείτε ως αυστριακή κυβέρνηση, αν δεν κάνετε τίποτα για το πι δέλτα πι, δεν θα πετύχετε τους στόχους σας ως υπουργό ε, Παιδείας. Σκεφτείτε το, προσπαθήστε να είστε κάπως ανοιχτός, γιατί αλλιώς είναι μειονέκτημα για τους νέους ε, στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Μα γιατί λέτε ότι δεν είναι σημαντικό αυτό για εμένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας παραπέμψω μόνο στο ότι το θέμα του ΠΔΠ είναι ζήτημα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και σας παρακαλώ να απευθυνθείτε εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά βεβαίως ε, και στο πλαίσιο των δικών σας αρμοδιοτήτων ε, έχετε κι εσείς κάποιες αρμοδιότητες. Αλλά πράγματι, ίσως ε, και οι Υπουργοί Οικονομικών θα έπρεπε να είναι κάπως πιο ανοιχτοχέριδες. Ε, Μαρίτερες Χιμένεθ. Sí, Ευχαριστώ πολύ. Η Αυστριακή Προεδρία, διαπιστώνω με τα χαράς, ενδιαφέρεται για την εκπαίδευση και την παιδεία. Και ευχαριστούμε για τη στήριξη που θέλετε να δώσετε στο Erasmus Συν. Ήμουν σκιώδη συγκίτρια για το θέμα αυτό και δεν θα επαναλάβω όλα τα σχετικά επιχειρήματα. Να σα επισημάνω απλώ ότι υπάρχουν πολλοί φοιτητέ που ακολουθούν ε, τον επιστημονικό κλάδο. Ε, είναι κάτι που το επιδιώκουν πολλοί στην Ευρώπη και το ζητούν, αλλά δυσκολεύονται να βρουν πανεπιστήμια ε, με υλικό και κύκλωμα θυμάτων εξειδικευμένο για να παρακολουθήσουν αλλού από τη σχολή τους ε, μέσω του Εράσμους. Εσείς τι μπορείτε να κάνετε για να διευκολύνετε τους φοιτητές που ενδιαφέρεται το Εράσμος. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ. Είπατε ότι οι φοιτητές δεν βρίσκουν το κατάλληλο πανεπιστήμιο. θα ήθελα κάποια στοιχεία εμπειρικά, γιατί δεν συμφωνώ. Ειδικά στις θετικές ε, επιστήμες έχουν μεγάλη κινητικότητα, οπότε νομίζω ότι ε, το βρίσκουν αυτό που θέλουν. Δεν μας ανησυχούν αυτές οι ειδικότητε γιατί μιλάνε ήδη διεθνείς γλώσσες όπως τα μαθηματικά. Αλλά μάλλον οι ανθρωπιστικές επιστήμες ε, μας ανησυχούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μπίλτ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε, που μας ε, Ευχαριστούμε, Υπουργέ, που μας θυμίσατε με την παρουσία σας σήμερα και συγχαρητήρια για αυτήν την εντυπωσιακή και αξιοσημείωτη έναρξη της Προεδρίας του Συμβουλίου. Η παρατηρήση μου σήμερα ε, αναφέρεται στο Εράσμους σε Η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει, γίνει, ε, έχει αποτελέσει αντικείμενο εγγύησης ως το 2020. Εδώ θα πρέπει να ανοίξουν νέε δυνατότητε συμμετοχή σε τρίτα μέρη αρκεί να σέβονται κάποιε προποθέσει και όρου, κυρίω ε, δημοσιονομικού και την λήψη αποφάσεων. Το κείμενο αυτό βρίσκεται ακόμη σε συζήτηση. Τι σκοπεύετε να κάνετε για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο Εράσμου Σύνδητο, είναι σημαντική χώρα υποδοχή για του Ευρωπαίου φοιτητέ. Οπότε η Βρετανική συνιστόσα του προγράμματο, εφόσον έλειπε, θα επέφερε σοβαρότατη βλάβη. Υπάρχει δυνατότητα ε, μάλιστα συμμετοχή τρίτων χωρών σε σχέση με το ισχύουν σήμερα για άλλα κράτη. Και αν ναι, ποια κράτη. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απολύτως μαζί σα. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πραγματικά πολύ αγαπητός προορισμός για τους φοιτητέ εράσμου και έχουμε και έναν οδικό χάρτη, ο οποίος ε, λέει, ω γνωστόν, ότι καταρχά πρέπει να τελειώσουμε με τον Brexit τη διαπραγματεύσει. Βέβαια, πρέπει πρώτα να συμβεί και μετά θα δούμε πώς θα δομηθούν οι σχέσεις μας. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει σχέση και μετά το Brexit, γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι απλώς δημοφιλής προορισμός, αλλά είναι πραγματικά εξαιρετική χώρα με πασίγνωστα πανεπιστήμια. Δεν θα μπορέσουμε να το διαπραγματευτούμε εμεί μέχρι να τελειώσει η Προεδρία μα δυστυχώ, αλλά εγώ ω Υπουργό Έρευνα και Εκπαίδευση σίγουρα θα φροντίσω να υπάρχει και μετά κάποια συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο και με τα υπόλοιπα κράτη βεβαίως, γιατί εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε τώρα τον εισηγητή μας που είναι υπεύθυνο για το Εράσμος. Ε, Ευχαριστώ, Υπουργέ, για την παρουσίασή σας και ευχαριστούμε που μας παρουσιάσατε τις προτεραιότητες της ε, Προεδρίας σας. Είμαι γείτον της χώρας σας, είμαι από τη Σλοβενία. Ε, χαίρομαι που έχετε συμπεριλάβει το Erasmus ΣΥΝ σε μια από τις προτεραιότητές σας ε, στο πρόγραμμα της Προεδρίας Στήριζετε την μεταρρύθμιση της διαδικασίας της Μπολόνιας και θέλετε να υπάρχει ένας ευρωπαϊκός χώρος της εκπαίδευσης και της ανώτατης στην Ευρώπη. Με χαροποιεί ιδιαιτέρως ότι έχετε ε, δώσει έμφαση στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση επίσης στην Ευρώπη. Και έχετε ιδιαίτερη γνώση του όλου ε, πεδίου αυτού. Είμαι βέβαιος ότι η Αυστριακή Προεδρία θα πετύχει πολλά. Ε, επειδή δεν υπάρχει πολλής χρόνος, έχω μία και μόνη ερώτηση. Μπορείτε να στηρίξετε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αλλάξει το όνομα του προγράμματος αυτού από το Εράσμους συν σε Εράσμους. Ευχαριστώ. Ähm, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε ικανοποιημένο με τις φιλοδοξίες μας. Για το συγκεκριμένο ερώτημα, για να ξαναγίνει το Erasmus ξανά Erasmus, Να σου πω, εγώ είμαι πλήρως ουδέτερος ως προς αυτό. Το σημαντικό είναι το Erasmus να διατηρηθεί ως όνομα. Γιατί είναι, αν θέλετε, ήδη ένα εμπορικό σήμα. Τώρα αν έχει συν, πλήν ή τίποτα μετά, εντάξει, εξαρτάται από εσάς. Ε, όχι μην, ναι, όχι πλήν, με συγχωρείτε, να έχετε δίκιο. Ναι, ναι, Άννα, έχουμε λεφτά, τα άλλα θα τα βρούμε. Έχω λοιπόν ακόμα πέντε ομιλητές. Και θα πρέπει να ακούσουμε και την κυρία Μπόγνερ Στράους. Λοιπόν, κοιτάξτε. Θα διακόψουμε εδώ και θα απαντήσουμε τις επόμενες ερωτήσεις στον επόμενο γύρο. Την επόμενη φορά. Ε, δεν ξέρω, μπορεί να κάνετε ερωτήσεις σε άλλους υπουργούς. Κυρία Μπόγνερ Στράους, έχετε τον λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πιο γρήγορα εγώ. Ε, ελπίζω να μην δυσαρεστήσω πάρα πολύ τους διερμηνείς. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα σας ε, παρουσιάσω τον τομέα της νεολαίας και τις προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας για τον ε, τομέα αυτό. Για μένα είναι πολύ σημαντικό η ε, νεολαία να ακουστεί. Πρέπει να ακούμε τους νέους μας, γιατί είναι το παρόν και το μέλλον μας. Οπότε πρέπει να τους δώσουμε ένα πλαίσιο, το καλύτερο δυνατό πλαίσιο, το οποίο μπορούμε να τους προσφέρουμε. Οι νέοι πρέπει να δημιουργήσουν την δική τους προσωπικότητα έτσι ώστε να μπορούν ως ενήλικες να μπουν στην κοινωνία και να προσφέρουν. Πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν για το μέλλον της κοινωνίας μας. Σύμφωνα με το Ευρωμαρόμετρο και μια ε, ε, έρευνα που έγινε, οι Ευρωπαίοι μεταξύ 15 και 30 ετών λένε ότι η πρώτη προτεραιότητα για αυτούς είναι η εκπαίδευση και οι δεξιότητες. Είναι καλό αυτό να τα ακούμε και με το πρόγραμμα Εράσμος νομίζω ότι έχουμε πραγματικά ένα πολύ επιτυχές παράδειγμα, όπως είπε ο συνάδελφος Φάσπαν, ένα εμπορικό σήμα, γιατί νομίζω ότι το, ο Εράσμος είναι αυτό ακριβώς οι νέοι μπορούν να μπουν στην Ευρώπη. Το Εράσμος είναι για τους ε, νέους. Είναι η πρώτη τους γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία, ενιαία. Πολλοί από αυτούς τους νέους συμμετέχουν και στην εθελοντική εργασία. Και αυτό απέρευσε ως αποτέλεσμα από την έρευνα. Έξι στους δέκα νέους έχουν ε, ε, πάρει μέρο σε τέτοια προγράμματα. Οπότε βλέπουμε ότι οι νέοι μα στην ε, Ευρώπη ασχολούνται και δραστηριοποιούνται πολύ. Υπάρχει μεγάλη παράδοση στην Ευρώπη σχετικά και έχουμε και την εθελοντική υπηρεσία πλέον. Οπότε θεωρώ ότι και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι πραγματικά μια σημαντική, ένα σημαντικό επίτευγμα, μια σημαντική κατάκτηση όπου οι νέοι μπορούν να μάθουν μπορούν να καταλάβουν την ένταξη, μπορούν να μάθουν την ανοχή και μπορούν να βγουν πιο δυνατοί από το πρόγραμμα αυτό, γιατί ακριβώς βρίσκονται εκεί για να υποστηρίξουν κάποιον. Κάνουν την εθελοντική τους εργασία για να μπορέσουν και οι ίδιοι να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική εμπειρία και η οποία τους ενισχύει και τους δυναμώνει. Γι' αυτό χαίρομαι που μέχρι το 2020 θα έχουμε 375 εκατομμύρια ευρώ και για, το, για τα έτη 2021 έως 2027 126 ε, εκατομμύρια ευρώ. Και 350.000 νέοι θα μπορέσουν να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν, να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα αυτό. Το έτος 2020 ε, λύγει το πρόγραμμα Erasmus+, το Erasmus το είπε και ο συνάδελφος Φάσμαν. Βεβαίως ε, το πρόγραμμα αυτό είναι ουσιώδου σημασίας και όσο όσο σε, όσο περισσότερους νέους μπορούμε να το προσφέρουμε, τόσο καλύτερα θα ενισχύσουμε και την ευρωπαϊκή κινητικότητα. Ε, μπορούμε δηλαδή ε, να προωθήσουμε 20 με 30% των συγκεκριμένων ετών και μια προσωπική άποψη. Όπως σε όλα τα project, σε όλα τα προγράμματα, θα έπρεπε να είναι πρόκληση αυτή για τους νέους ή για ομάδες νέων να μπορούν να πάρουν μέρος σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και γι' αυτό και εδώ ισχύει το ότι πρέπει να βάλουμε ένα λιθαράκι για να μπορέσουμε να σπρώξουμε στους νέους τα προγράμματα αυτά. Από την άλλη πρέπει να πούμε ξεκάθαρα και ήδη αναφέρθηκε ο συνάδελφος ότι το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να γίνει λιγότερο γραφειοκρατικό και θα πρέπει να χαμηλώσει και το ε, όριο για τη συμμετοχή. Είναι σημαντικό αυτό για τους νέους να μπορούν να μπαίνουν πιο εύκολα στο πρόγραμμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και νέους που βρίσκονται πιο μακριά από το χώρο της εκπαίδευσης, να διευκολύνουμε τα πράγματα και ακόμη και στην διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων. Για τον τομέα της νεολαίας, από το Erasmus ε, Συν, περιμένουμε 3,1 δις ευρώ. Ωραία τα κονδύλια αυτά για να μπορέσουν να αναπτυχθούν περαιτέρω οι νέοι Μιλούμε για 30 δις συνολικά και όπως είπα πάντα μπορούμε να ζητούμε λίγο παραπάνω αλλά οι νέοι ήδη θα μπορούν να βλέπουν ως πρόκληση αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσουν να κάνουν τις αιτήσει τους. Και βεβαίως θα πρέπει να διατηρήσουμε και ένα πλαίσιο ποιότητας και προϋποθέσεων. Μετά, η στρατηγική για την νεολαία. Χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική για την νεολαία. Υπάρχει η σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιπλέον μέσω ε, ενοποίησης διαφόρων ε, προγραμμάτων ε, συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα στην Σόφια αρκετές χιλιάδες νέοι. Παρουσιάστηκαν οι 11 στόχοι για την νεολαία που νομίζω ότι περιλαμβάνουν τα πάντα όσα ευχόμαστε για τους νέους. Και αυτό είναι δική μου ευχή επίσης να γίνουν τα πράγματα λίγο πιο συγκεκριμένα. Οι νέοι και ο χρόνος είναι πραγματικά δραστική η αλλαγή. Τα πράγματα αλλάζουν τόσο γρήγορα και εμείς πρέπει να τα παρακολουθούμε. Οι νέοι το ξέρουν αυτό πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό εγώ τους είμαι ευγνώμων που έθεσαν αυτούς τους 11 στόχους και βεβαίως θα προσπαθήσουμε κι εμείς στο βαθμό που μπορούμε να τους ενσωματώσουμε στην νέα στρατηγική για την νεολαία. Χαίρομαι λοιπόν ως Προεδρεύουσα του Συμβουλίου που μπορώ να ενισχύσω την ε, πολιτική για την νεολαία τους επόμενους έξι μήνες και να τη φέρουμε πιο κοντά στους νέους. Και εσείς φυσικά είσαστε σημαντικός εταίρος μας και είναι σημαντικό εδώ να πω ότι πρέπει να ενισχύσουμε το διάλογο με τα θεσμικά όργανα, αλλά πρέπει να ακούσουμε και τους νέους μας. Οι νέοι μας είναι το μέλλον μας. Και ελπίζω ότι ως προς αυτό θα συμφωνήσετε μαζί μου. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν χρησιμοποιήσατε και τα 10 λεπτά που σας έδωσα. Ε, σας ευχαριστώ. Να ε, ξεκινήσουμε με τους ε, συναδέλφους που είχαν, δηλώσει, που είχαν ζητήσει το λόγο για τον προηγούμενο γύρο και να θέσουμε τα ερωτήματα στην Υπουργό. Η κυρία Μπόσκουβα έχει το λόγο. szépen miniszternek Ευχαριστώ, Υπουργέ, για τις παρουσιάσεις σας. Είναι μεγάλη μου, ε, με μεγάλη ικανοποίησή σας άκουσα να αναφέρετε ε, πολλά από τις προτεραιότητες της Επιτροπής μας, μεταξύ των οποίων το Εράσμος είναι η εκμάθηση γλωσσών και άλλα μεταξύ των προτεραιοτήτων σας. καθώς και την αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων. Θέλω να τονίσω το εξή. Ε, εγκρίναμε έκθεση για τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευση και θα ήθελα να την θυμίσω και να σας επισημάνω την έκθεση αυτή. Υπήρχαν πολλές σημαντικές παρατηρήσεις εκεί για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεχομένως και εκτός Ένωσης. Υπάρχουν πολλές σημαντικές συμβουλές λοιπόν σε αυτή την έκθεση και καλό θα ήταν να δούμε όχι μόνο το επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και παρακάτω. Όσο πιο νωρίς ένα παιδί ε, μπει στο εκπαιδευτικό σύστημα, τόσο περισσότερο έχει πιθανότητες να παραμείνει σε αυτό και μετά να είναι και επιτυχές στην αγορά εργασίας. Οπότε, ξέρω ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αποφασίσουν πόσο θα δαπανίσουν ε, στις πολιτικές παιδείας τους. Όμως εγώ ήθελα να σας ζητήσω να ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη να δαπανούν περισσότερα και να βελτιώνουν την ποιότητα των ε, εκπαιδευτικών του ιδρυμάτων. Είναι σημαντικό αυτό για την ε, ένταξη και για τα παιδιά που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι θα μπορέσετε να καταγράψετε όλα όσα αναφέρουν οι συνάδελφοι. Ε, όχι, όχι, ο, ο συνάδελφος πίσω από εσά και μετά εσείς. Thank you. Uh, it was certainly very... Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας, Υπουργέ. Κυρίως καλωσορίζω το γεγονός ότι αναφερθήκατε στους νέους ε, ως το παρόν και το μέλλον. Κάποιοι ε, τους αναφέρουν μόνο ως κάτι μελλοντικό. Ξεχνάμε ότι αποτελούν μέρος του παρόντος. Αυτό είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Ένα συγκεκριμένο θέμα που σχετίζεται και με το Εράσμος που έχει ε, αναφερθεί τόσες φορές και στις δικές σας παρουσιάσεις. Είναι μια νέα πρωτοβουλία που απευθύνεται ιδιαίτερα στους νέους. Αυτή που ονομάζεται Discovery EU ή τέλος πάντων το σύστημα Interrail το εισιτήριο Intel βλέπετε είναι ένα πρόγραμμα ε, που αναπτύσσεται. Ε, πρώτα ήταν σε πειραματικό στάδιο, τώρα θέλουμε να γίνει μόνιμο. Τα πορίσματα, η αντιδράση των νέων και το feedback που είχαμε ήταν πολύ θετικό για του νέου και φοιτητέ. Και η ερώτηση είναι αν θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε ως ένα ξεχωριστό πρόγραμμα, ε, αυτόνομο από το Ε, Και πώ θα χρηματοδοτηθεί. ένα άλλο χώρο που είναι ζωτικό, είναι αυτό τη εθελοντική εργασίας. Ε, πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να ενθαρρύνουμε τον εθελοντισμό των νέων να συμμετέχουν σε με κυβερνητικέ οργανώσεις, στο Σώμα και σε άλλα. Και τέλος, καλωσορίζω την μνήμα σας στους νέους που δεν έχουν οργανωθεί κάπως πολιτικά, ε, δεν βρίσκονται σε κάποια ένωση, κίνημα, ε, φοιτητικό κόμμα κτλ. Αλλά υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς θα φτάσουμε σε αυτούς, με τι επικοινωνιακή πολιτική. Δεν πρέπει να σκεφτούμε τους νέες, τις νέες μορφές και την πραγματικότητα της επικοινωνίας. Είναι σημαντική αυτή η διάσταση, διότι η πλειοψηφία των νέων κάπως θα περιθωριοποιηθούν, διότι η επικοινωνική μας πολιτική δεν φτάνει ως τα αυτιά τους. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις ε, και τις ερωτήσεις σας. Όσον αφορά το Discover, υπάρχει μια πρόταση προϋπολογισμού 700 εκατομμυρίων ευρώ από το 2021 μέχρι το 2027. Αυτή την στιγμή νομίζω το βλέπουμε παρά το ότι υπάρχει αυτό το θέμα του Interrail που αναρωτιόμαστε τι σχέση έχει με την μάθηση. Αλλά όσοι ταξιδεύουν ε, μαθαίνουν. Για μένα το Interrail ήταν η πρώτη μου εμπειρία και ταξίδι στο εξωτερικό και έμαθα πάρα πολλά ε, πράγματα. Αυτήν τη στιγμή ήδη 100.000 νέοι έχουν ενδιαφερθεί για αυτό. Για 15.000 ε, υπήρχαν ειστήρια. Ταξιδεύουν αυτοί ήδη και 700 εκατομμύρια ευρώ νομίζω είναι ε, ο προτινόμενος προϋπολογισμός για να διατηρηθεί. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είπα ήδη ότι για εμένα είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Νέοι οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά στην Ευρώπη να βοηθήσουν αυτό βεβαίω δεν μπορούμε παρά να το υποστηρίξουμε και έχει πολύ ψηλή προτεραιότητα για την Αυστριακή Προεδρία αυτό το νομοθετήμα και το 1 δισεκατομμύριο και κάτι ε, έχουν προβλεφθεί για 30.000 νέους. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο το οποίο προβλέπεται και θα στηρίξει αρκετούς ε, νέους. Εγώ θα ήθελα βέβαια να έχει ένα χαμηλότερο κατόφλι, να είναι λιγότερο γραφειοκρατικό, μιλώντας για τη χώρα μου δηλαδή. Είναι και κάπως δύσκολο για τους νέους ε, να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα και νομίζω ότι κάτι θα κάνουμε στην διευκόλυνση. Όσον αφορά την επικοινωνία είμαι πλήρως στο πλευρό σας. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες επικοινωνίας για να ακούσουμε τους ε, νέους. Και έχοντα τώρα ακριβώς αυτούς 50.000 νέους ε, που ρωτήσαμε εν ώψη της Προεδρίας, της Τριπλής Προεδρίας, θα έλεγα ότι το εκμεταλλευτήκαμε, εκμεταλλευτήκαμε τα νέα κοινωνικά μέσα. Βεβαίως, εντάξει, παντού υπάρχουν κενά, δεν υπάρχουν παντού τα κοινωνικά μέσα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντα κατά νου και να ακούμε τους νέους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ όμως όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Νέκο. Σας ευχαριστώ και καλή σας μέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερος για το ότι μιλάμε για τις δικές σας πολιτικές προτεραιότητες. Αυτό το οποίο δεν άκουσα είναι το πρόβλημα της ανεργίας και των νέων. Είναι ένα πρόβλημα στο οποίο εργαζόμαστε εδώ και καιρό, αλλά βεβαίως εξακολουθεί να υπάρχει, ειδικά ε, στα άτομα εκείνα τα οποία δεν εκπαιδεύονται και δεν ε, εργάζονται. Γι' αυτό θεωρώ ότι ακριβώς αυτό το πρόβλημα πρέπει πρώτα απ' όλα να αναγνωριστεί. Γι' αυτό ακριβώς ε, πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες στους νέους. Αλλιώς θα έχουμε την πρώτη γενιά η οποία θα είναι φτωχότερη από τους γονείς της. Ε, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτησή σας. Ναι, να αναφερθώ στο θέμα της ενέργειας των νέων. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους στην Ευρώπη, κάποιες χώρες περισσότερο, κάποιες χώρες λιγότερο. Στην Αυστρία έχουμε την ευτυχία να έχουμε σχετικά χαμηλή ανεργία των νέων, γύρω στο 9%, αλλά ελπίζω με το Ευρωπαϊκό Σώμα σε ένα κόμμα, ε, κομμάτι με συγχωρείτε, του προπολογισμού να πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Το βλέπω θετικά και αρνητικά με την έννοια ότι θα δώσουμε ε, κάποιες δουλειές ή πρακτικές ασκήσεις που θα διαρκούν τουλάχιστον τρεις μήνες, αλλά βεβαίως υπάρχει και η θλιβερή πτυχή ότι δεν ε, εκμεταλλευόμαστε πλήρως, θα έλεγα, τους νέους σε δουλειές και πρακτικές ασκήσεις όπου είναι πολύ περιορισμένη η αμοιβή. Δηλαδή, αφενός, εντάξει, είναι θετικό, από την άλλη είναι αρνητικό. Γι' αυτό ακριβώς το ήθελαν αυτό τόσες πολλές ε, χώρες, ε, αλλά έχουν τελείως διαφορετικές αντιλήψεις, γιατί έχουν και διαφορετική ανεργία των νέων. Έχουμε όμως μια ευκαιρία εδώ πέρα με την ε, ψηφιοποίηση. Και ακριβώς αυτό είναι το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Και να δούμε ακριβώς το θέμα της εκπαίδευσης και μάλιστα πριν από το σχολείο την ε, στοιχειώδη εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω τσεχικά. Και θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα και στους δύο υπουργούς. Ε, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ καταρχάς για την ε, σαφή θέση που πήρατε για το θέμα της νεολαίας θα ήθελα να μιλήσω για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Να, θα έπρεπε το Συμβούλιο να ασχοληθεί παρόλο που το, με το θέμα αυτό, παρόλο που το Κοινοβούλιο είναι ακόμα σε διαδικασία συνδιαλλαγή. Έχουμε την ολοκλήρωση του τριμερούς διαλόγου για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Το στηρίξαμε, το βασίσαμε σε εμπειρίες κτλ. Και προετοιμάζεται κάτι για, τις επόμενες, για την επόμενη ε, περίοδο, για την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Και είναι σημαντικό και εσεί από τη δική σα τη μεριά στο Συμβούλιο να υποστηρίξετε την κατεύθυνση που έχουμε λάβει σε αυτή την περίοδο. Για την ε, υπηρεσία, ας πούμε, θελοντικής εργασίας κλπ και μετά βεβαίως να γίνουν και τα υπόλοιπα βήματα. Και φυσικά εμείς χαιρόμαστε πολύ για την ε, συνεργασία. Και για τον Υπουργό Παιδείας θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε την δυνατότητα της αναγνώρισης των ε, διπλωμάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γιατί εμείς ασχολούμαστε με το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης ε, της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κυρίως μιλώ και για την αυτόματη αναγνώριση. Υπάρχει μια διαφορά με την ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν έχουμε τόσο δομημένη, ας πούμε, ε, διαδικασία. Δεν υπάρχουν δηλαδή οι απαραίτητε δομές για να γίνει αυτό. Τι δυνατότητες βλέπετε να υπάρξει όντως αναγνώριση για την δευτεροβαθμία εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, παρακαλώ και εσά να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ. Καταρχάς να ευχαριστήσω την, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που τα κατάφερε τόσο καλά και έθεσε το σημείο κίνησης για τις μελλοντικέ διαπραγματεύσεις που είναι βεβαίως η συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Κομισιόν, που είναι η συμφωνία της 27ης Ιουνίου, ο Υπουργός Φάσμαν θα μπορούσα να σας δώσω μία πολύ μακρά απάντηση, κυρία Νέκοφ, για την ε, ε, ανεργία των νέων, αλλά δυστυχώς δεν με αφήνει να κάνω διάλεξη, κυρία Πρόεδρος. Για την ε, κυρία Σέντροβα. Ε, αναγνώριση, η αναγνώριση των πανεπιστημίων, των διπλωμάτων των πανεπιστημίων λειτουργεί. πρέπει να έχουμε μία δεσμευτική και συγκρίσιμη διαδικασία ποιοτική αξιολόγηση. Για τα δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά εκεί πρέπει να φτάσουμε. Πρέπει να έχουμε διαφανεί διαδικασίε, ε, ποιοτικά μέσα και για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτό είναι η μόνη δυνατότητα που έχουμε ώστε να καταλήξουμε σε δεσμευτική ε, αναγνώριση των διπλωμάτων της δευτεροβάθμιας. Ευχαριστώ οι επόμενοι ε, υπουργοί περιμένουν στην πόρτα. Οπότε τα υπόλοιπα τέσσερα άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο να ε, συγχωνεύσουμε λίγο τις παρεμβάσεις τους και να πάμε στο επόμενο σημείο. Τζότο, Βερ, Κώστα και κυρία Τρούπελ. Ε, ένα λεπτό καθένα σας και όχι παραπάνω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος, ο κύριος Σερνατζότο. Αγαπητοί Υπουργοί, ε, πραγματικά είναι αξιοσημείωτες οι προτεραιότητες που έχετε θέσει, αναγνώριση των δεξιοτήτων, ε, ε, η χρήση όρων που χρησιμοποιούν, χρησιμοποιούμε εμείς αλλά όχι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. τους επόμενους 6 όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν τελικά σε μια διαφορετική πολιτική για την επικοινωνία σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Έχουμε αρκετά αντιφατικές συζητήσεις για την αναγνώριση των δεξιοτήτων κτλ. Στις, στην ομιλία σας το αναφέρατε αυτό ξεκάθαρα και νομίζω ότι θα μπορούσαμε όντως να βοηθήσουμε την Ευρώπη αν κάναμε κάτι τέτοιο. Αυτή νομίζω είναι η πιο σημαντική και η μόνη επιτάχυνση που θα βοηθούσε είναι σημαντικό για τη δόμηση της ε, Ευρώπης, αν όντω επιταχύνουμε στον τομέα της εκπαίδευση. Ωραία, η κυρία Κώστα, γιατί ο άλλος ομιλητής ε, αποχώρησε. Ναι, ναι, τρία πράγματα μόνο και δεν θα κάνω σχόλια. Πρώτον, είδα στις προτεραιότητές σας κάτι το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Λέτε κάποια πράγματα για τον ρόλο στην εργασία των ε, νέων μεταναστών ε, και προσφύγων. Με ενδιαφέρει να καταλάβω λίγο καλύτερα εδώ πέρα τι εννοείται. Δεύτερον, ε, μιλάτε ακριβώς ε, όχι το τι θα γίνει μόνο με το νέο πρόγραμμα, αλλά και το σχέδιο εργασίας για το 19 και το 20 για τη στρατηγική για τους νέους. Αν θέλετε να μου εξηγήσετε και εδώ πέρα τι σκοπεύετε να κάνετε για την πολιτική για τους νέους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Υπουργέ, περιμένετε. Περιμένετε να ακούσουμε άλλη μια ερώτηση και μετά θα απαντήσετε. Χέλγα Τρούπελ, θα επανέλθω στο θέμα των μειονεκτικών νέων που στις μεγάλες πόλεις, αλλά ειδικά στην Ήπεθρο, έχουμε και για να έχουν ίσες ευκαιρίες θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική οποία ε, θα πρέπει να πηγαίνει και προς την κατεύθυνση αυτή που έχουμε με το Ευρωπαϊκό Σώμα Θα λοιπόν να μάθω τι προθέσεις έχετε ως Προεδρία. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, θα προσπαθήσω λοιπόν να απαντήσω σύντομα. Κυρία Κώστα, για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου έχουν ως εξής η απάντηση είναι ναι. Για τη στρατηγική για τους νέους η απάντηση είναι επίσης ναι. Για το επόμενο εξάμεινο ε, θα έχουμε ένα άτυπο Συμβούλιο Νεολαίας το Σεπτέμβριο στην Βιέννη με υπουργού, ε, με ειδικού, με ΜΚΟ και με βουλευτές βεβαίως, ευρωβουλευτές. Να δούμε αν θα επεξεργαστούμε μια τη στρατηγική και να δούμε πώς θα την εφαρμόσουμε γιατί έχουμε μέχρι στιγμής ε, προγράμματα που καλύπτουν μόνο τρία έτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ναι. Κύριε ότι μιλήσατε για κάποιες ε, συζητήσεις που θα πρέπει να γίνουν για την αναγνώριση ευρωπαϊκών ε, πανεπιστημίων και προγραμμάτων. Εντάξει, όλου αρέσουν επίμαχοι συζητήσει, αλλά είστε σίγουρο ότι θέλετε να γίνουν στο Συμβούλιο. Ναι. Κυρία Τρίπελ, ε, είναι σοβαρό το θέμα το οποίο αναφέρατε ε, και πραγματικά το έχω σκεφτείτε ότι μπορούμε να κάνουμε. Από τον τομέα της εκπαίδευσης, μιλώντας μόνο, ένα από τα μέτρα είναι οπωσδήποτε το θέμα της διπλής Εκπαίδευση που έχουμε σε Ελβετία, Αυστρία και Γερμανία ε, που ίσως είναι ενδιαφέρον για άλλες χώρες. Γιατί ακριβώς αυτοί, αυτές οι δύο κατευθύνσεις που έχουμε αφενός ε, την θεωρητική εκπαίδευση στο σχολείο και την πρακτική εκπαίδευση μετά ε, για την αγορά εργασίας για να μπαίνουν σε μια δουλειά οι μαθητές έχει οδηγήσει σε μεγάλα ποσοστά επιτυχίας, απασχόλησης δηλαδή. Οπότε ακριβώ το θέμα της εκπαίδευσης και κατάρτισης ε, της επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ένα θέμα προτεραιότητας γιατί είναι καλό μέσο καταπολέμησης της ανεργία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει η Πρόεδρος, παρατηρούμε λοιπόν από τις ε, ερωτήσεις και τη διάθεση των συναδέλφων πως είναι θέματα που μας απασχολούν. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που ήσασταν στην διάθεσή μας και περισσότερο από όσο προβλεπόταν. Ε, δυστυχώς τώρα πρέπει να διακόψουμε γιατί οι συνάδελφοι είναι εδώ πέρα έξω από την πόρτα. Οπότε δεν γίνει τέλειος. Λοιπόν, τους επόμενους έξι μήνες οπωσδήποτε θα είμαστε σε επαφή. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν ε, πάρα πολύ και καλή επιτυχία στην Προεδρία σας. So, Αγαπητοί συνάδελφοι, ερχόμαστε στο δεύτερο κομμάτι της πρωινής μας συνεδρίασης και χαίρομαι πολύ που μπορώ να καλωσορίσω μετά την ε, πρώτη επιτυχή ανταλλαγή απόψεων με τους δύο συναδέλφους τους και τον ε, κύριο Μπλούμελ και τον κύριο Στράχε. Ε, βλέπετε ότι πήρε λίγο παραπάνω η συζήτηση, αλλά το θέμα της εκπαίδευσης ε, πραγματικά συγκινεί πολύ την ε, Επιτροπή μας. Τώρα βρισκόμαστε στον, στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού. Χαίρομαι λοιπόν που μπορούμε να καλωσορίσουμε τον αντικαγκελάριο κύριο Hans Christian Strache, είναι υπεύθυνο υπουργό για τον αθλητισμό και τον κύριο Γκέρνοτ Μπλούμελ, ο οποίος είναι υπουργό τέχνης, πολιτισμού και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχουμε συμφωνήσει ότι ο καθένας σας θα πάρει 10 λεπτά για την εισαγωγική σας παρέμβαση. Ε, θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Μπλούμελ, 10 λεπτά και μετά θα κάνουμε ένα πινκ-πονκ ερώτηση-απάντηση, ερώτηση-απάντηση. Μην ανησυχείτε. Είμαστε πολύ τυπικοί ε, ε, επιτροπή και θα, θα τους προλάβουμε όλου. όλους. Και μάλιστα αρέσει και στα μέλη το ping-pong. Γίνονται τα πράγματα λίγο πιο ενδιαφέροντα. Κύριε Μπλούμελ, καλώς ήρθατε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κύριε Αντικακυλάρη. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Καταρχάς, να πω ότι γνωρίζω το Κοινοβούλιο δεν ήμουνα πολύ ενεργός ε, έτσι ως δραστηριοποιούμενος, αλλά έκανα δύο φορές πρακτική στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πραγματικά α, ε, χαίρομαι που τώρα μπορώ να έχω έναν επίσημο τίτλο και μια επίσημη θέση και να σας μιλώ από εδώ. Καταρχάς να μιλήσω για τις βασικές ε, προϋποθέσεις πλαίσιο για την Προεδρία μας. Είναι η τρίτη φορά που η Αυστρία από το 1998 και το 2006 αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου και η Προεδρία αυτή βεβαίως ε, αντιμετωπίζει πάρα πολλές προκλήσεις. Ξέρουμε όλοι ότι από τη μια έχουμε το θέμα της μεταναστευτικής κρίσης, έχουμε το Brexit, έχουμε άλλα θέματα που είναι επίγοντα και γι' αυτό σκεφτήκαμε ποιο, είναι το, ποιο θα πρέπει να είναι το μότο της Αυστριακή Προεδρίας και αποφασίσαμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι η Ευρώπη που προστατεύει. Προστασία τη ενία βέβαια. Προστασία από την παράνομη μετανάστευση, αλλά προστασία και τη ευημερία μας. Εμβάθυνση τη εσωτερική αγοράς και προστασία της σταθερότητας στην γειτονιά μα. Να δούμε δηλαδή αν θέλουμε να εξάγουμε σταθερότητα ή αν θέλουμε να εισάγουμε αστάθεια. Αυτά κυρίω αφορούν τι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη και των Δυτικών Βαλκανίων. Επίση, ένα σημαντικό θέμα τη Προεδρία μα είναι το θέμα της επικουρικότητας. Σημαντικό θέμα, τεράστιο θέμα, όλοι είναι υπέρ, αρκεί να μπορέσουμε να ορίσουμε τι σημαίνει η επικουρικότητα. Εκεί όταν πάμε να το ορίσουμε πιο συγκεκριμένα, τα πράγματα αλλάζουν. Και ο Επίτροπος Τίμερμανς έκανε πραγματικά μια σημαντική παρέμβαση για να εξεύρουμε ε, σαφήνεια ως προς αυτό και θα υπάρξει και η αντίστοιχη διάσκεψη στην Αυστρία για να αφοσιωθούμε στο θέμα αυτό ακριβώς. Γενικώ ε, για τα θέματα που θα, ε, με τα οποία θα ασχοληθεί η Προεδρία μας, Έχουμε τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τα οποία δίνουν μια νέα κατεύθυνση στην συζήτηση για τη μετανάστευση στην Ευρώπη και θέλουμε τα συμπεράσματα αυτά να τα προωθήσουμε και κατά τη διάρκεια της δικής μας Προεδρίας. Κυρίως για την άτυπη συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στις 20 Σεπτεμβρίου στο Ζάλτσμπουργκ. Θέμα ευημερία ανταγωνιστικότητα εκεί κυρίως θα ασχοληθούμε με την ψηφιακή οικονομία. Είναι μεγάλη πρόκληση για το πώς μπορούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο ψηφιακό χώρο να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να έχουν κέρδος. Όχι μόνο ε, οι μεγάλοι γίγαντες του ε, ε, διαδικτύου, αλλά να υπάρχει και μια ισότητα όπλων για όλους. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα όπου και τα τρία θεσμικά όργανα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για το πώς θα κινηθούμε. Τώρα, προοπτικές για τα κράτη για, τις, ε, για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, στο θέμα αυτό θα, με το θέμα αυτό ασχολήθηκε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και καταλήξαν σε ένα συμβιβασμό όπου υπάρχει σαφή πρόθεση για τα ε, ένταξης για τα κράτη των ε, Δυτικών Βαλκανίων. Οι προσπάθειες που γίνονται στι χώρε αυτές, α πούμε το, η επίλυση του ονοματολογικού στην ΦΥΡΟΜ, είναι σημαντικές ε, προσπάθειες. Εντάξει. Συνολικά λοιπόν υπάρχουν κάποιες προκλήσεις ε, τις οποίες πρέπει να ομαδοποιήσουμε. Έχουμε και το θέμα του Brexit. Αυτή την εβδομάδα είδαμε ότι ε, το Ηνωμένο Βασίλειο έβαλε την δική του γραμμή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι τεράστια η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με το Brexit και σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και με τις διαπραγματεύσεις για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας ε, παρουσιάσουμε τις γενικές προτεραιότητες του, της Προεδρίας μας. Αλλά εγώ θέλω να επικεντρωθώ και στα, κυρίως στα θέματα του πολιτισμού. Το Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού θα γίνει στις 27 ε, Νοεμβρίου και η ε, Αυστριακή Προεδρία θα ασχοληθεί με τέσσερα βασικά θέματα ως προς αυτό. Καταρχάς, έχουμε το θέμα του μέλλοντος του πολιτισμού, των δημιουργικών ε, τεχνολογιών και του ψηφιακού χώρου στο μέλλον θα είναι δυνατόν να έχουμε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα, κυρίως για τους ε, πολιτιστικούς ε, φορείς, μόνο εάν αυτοί οι πολιτιστικοί φορείς που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να, κερδίσουν να και κάποια χρήματα. Αν τα χρήματα πάνε μόνο προς τη ΣΥΠΑ, Και αν τελικά έχουμε ένα, ε, μια ισότητα όπλων που δεν συμβαίνει τώρα, τα πράγματα θα βελτιωθούν. Επίσης, έχουμε το νέο ΠΔΠ για τη Δημιουργική Ευρώπη, 21-27. Ε, σε, σε επίπεδο Συμβουλίου θα το προωθήσουμε αυτό. Τρίτο σημείο, η ψήφιση του επόμενου πολιετούς ε, σχεδίου για τον πολιτισμό για μετά το 2019 που επίσης θα ασχοληθεί και με, την νέα, με τον θεματολόγιο και τον πολιτισμό. Και τέταρτον, μία προτεραιότητα για, τον, για, την Ευρωπαϊ... για το έτος Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018. Επίσης, ε, θα έχουμε ένα, ένα πρόγραμμα πλαίσιο πολύ φιλόδοξο και ενδιαφέρον. Θα δημιουργήσουμε από τη μία, μία ε, γέφυρα μεταξύ καινοτομίας ε, και πολιτισμού, όχι όμως μόνο στα πλαίσια που, έχουμε, που τα έχουμε εδώ. Έχετε ακούσει σε πολλά σημεία να παίζει μουσική παραδοσιακή, ε, βιενέζικη. Ε, έχουμε διάφορα είδη μουσική τα οποία ε, ακούμε κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας μας. προσπαθούμε να φέρουμε τους πολίτες και εμάς, τους ίδιους, σε επαφή με τα διάφορα είδη μουσικής στα πλαίσια του πολιτισμού. Και σήμερα θα ανοίξουμε άλλη μια ε, έκθεση εδώ στο Κοινοβούλιο για το θέμα της διαχείρισης των ΜΜΕ ε, στα πλαίσια του πολιτισμού. Η ε, Προεδρία μας θα κάνει μια σημαντική συζήτηση για τον δημιουργικό τομέα. Και βεβαίως εδώ μιλούμε κυρίως για το θέμα του τι γίνεται μελλοντικά με τις online πλατφόρμες. Οι συνθήκες ανταγωνισμού ήδη αναφέρθηκαν. Είναι μία από τις βασικές πτυχές, έτσι ώστε δημιουργική, ε, ε, ο δημιουργικός τομέας να μπορεί να είναι επιλέξιμος για χρηματοδότηση. Υπάρχουν διάφορες ε, προϋποθέσεις αλλά η, ο τομέας της μουσικής, η βιομηχανία της μουσικής ε, θα αναδομηθεί για να, δει, για να δούμε τι γίνεται με τα εισοδήματα και, την, και το κέρδος. Εγώ ας πούμε από το 90 με το χαρτζελίκι μου έπαιρνα CD και μετά ξαφνικά ε, ε, τα ανταλλάσαμε, Τέλο τέλος πάντων εντάξει δεν θα μπω σε λεπτομέρειες και κάποια στιγμή τα πράγματα έγιναν πολύ πιο απλά όλα τα έχουμε ε, στο τηλέφωνό μας. Ε, πατάμε ένα κουμπί, πληρώνουμε για τη μουσική και παίρνουμε τη μουσική που θέλουμε. Αλλά επειδή γίνεται αυτό και το τομέα τη μουσική, μπορεί να γίνει και για άλλους δημιουργικούς τομείς. Οπότε το θέμα είναι πώς θα καταφέρουμε οι ε, ιδιοκτήτες της πνευματική ιδιοκτησία να μπορούν να έχουν ε, εισόδημα για τα ε, έργα τους. Θα πρέπει λοιπόν και στον ψηφιακό χώρο να υπάρχει μια προστασία της πνευματική ιδιοκτησίας. Αυτό δεν ισχύει προς το παρόν για την για τον ψηφιακό χώρο ή θα πρέπει να ισχύει η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας για όλα ή για τίποτα. Μετά έχουμε τη διάσκεψη ακριβώς για το θέμα αυτό που θα γίνει στην ε, Βιέννη. Για το περιεχόμενο του ψηφιακού χώρου. Εκεί θα κάνουμε την ε, συζήτηση για, με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Για την Δημιουργική Ευρώπη τώρα και το σχετικό πρόγραμμα. Χαιρετίζουμε το ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ανεξάρτητο και ε, μπορεί να προωθηθεί από την Κομισιόν. Ο τομέας πολιτισμού και δημιουργικού θα είναι σημαντικός για την ε, κοινωνία και για την ε, οικονομική απόδοση. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή απάντηση απέναντι στα ερωτήματα που τίθενται. Αυτό που δεν θέλω να ξεχάσω είναι οι διαπραγματεύσεις για το φιλόδοξο πρόγραμμα, οι οποίε βεβαίω θα εξαρτηθούν από τις συζήτησει που θα γίνουν για τι ε, δημοσιονομικέ προοπτικέ 2021-2027. Τρίτο σημείο για το θεματολόγιο για τον πολιτισμό και το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2019 συν. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει την ε, νέα, το νέο θεματολόγιο για τον πολιτισμό και εκεί υπάρχουν ε, απαιτήσει από το Συμβούλιο για την στενότερη συνεργασία. Υπάρχουν διάφορες ε, πτυχές ε, που επίσης θα παίξουν ρόλο και εμείς κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα φροντίσουμε να τις προωθήσουμε. Ε, για το έτος τώρα της πολιτιστικής κληρονομιάς, ξέρουμε ότι είναι ένα θέμα σημαντικό και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό, γιατί μας δίνει και την ευκαιρία να ερμηνεύσουμε το θέμα αυτό εντός συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα και πρέπει νομίζω να καταλάβουμε ε, τι είναι η πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη. Γιατί μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα τα οποία συζητούμε. Μιλάμε πάντα για διάφορες αντικρουόμενες απόψεις, αλλά πρέπει να δούμε τι είναι κοινό στην Ευρώπη. Τι είναι αυτό που ορίζει την ευρωπαϊκή ταυτότητα αν υπάρχει κάποιος τομέας ο οποίος, υπάρχουν, ο οποίος διέπεται και από διαφορές αλλά και από ομοιότητες και που αυτά μπορεί να βοηθήσουν να βελτιωθεί, είναι σίγουρα ο τομέας της, του πολιτισμού και της τέχνης. Οπότε αυτό είναι μια διαδικασία ε, ε συνειδητή που πρέπει να γίνει. Η ποικιλία που υπάρχει στον πολιτισμό είναι σημειοθετικό. Γι' αυτό και εμεί και στη Βιέννη αλλά και σε όλη την ε, ε, ε, Βιέννη δίνουμε μεγάλη σημασία στην στην, στον πολιτισμό και στο εκτήριο του Συμβουλίου υπάρχει το πρόγραμμα ε, ε, τέχνη, το, το ε, Museum in a Nutshell, ένα μουσείο ε, μικρό το οποίο μπορείτε να το, να το δείτε. Υπάρχει επίσης μια διάσκεψη το Europe for Culture 6 και 7 Δεκεμβρίου στη Βιέννη. Και εκεί επίσης ε, θα φροντίσουμε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν πολύ εντατικό εξάμεινο. Ε, ξέρω ότι έχω ξεπεράσει το χρόνο μου, γι' αυτό κλείνω. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και βεβαίως περιμένω τα ερωτήματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Και περνάμε τώρα στις ερωτήσεις. Ε, σας παρακαλώ να είστε σύντομοι για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε στην ώρα μας. και μην σπαταλάμε χρόνο. Η κυρία Φερχάιν. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα. Χάρηκα για αυτό το οποίο είπατε. Ποικιλομορφία και ενότητα. Νομίζω πως είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Ιδιαίτερα στον πολιτισμό, ενδεί τον πολιτισμό θα δει ε, πως υπάρχουν οι διάφορες επιρροές ε, ε, διάφορες περιοχές που οδήγησαν στο δικό μας πολιτισμό χωρίς Ρωμαίους δεν θα είχαμε και την Καθολική Εκκλησία το γοτθικο ρυθμό τους Γάλλους από την άλλη Οπότε είπα, είχαν πάντα αμοιβέ επιρροές στην Ευρώπη. Λοιπόν, αναφέρατε κάτι το σημαντικό για τον δημιουργικό τον τομέα, τον οποίο εάν ναι, θέλουμε να ενισχύσουμε θα πρέπει να ισχύσουν οι κανόνες που είχαμε στον αναλογικό κόσμο και στον ψηφιακό κόσμο. Ξέρετε πως εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια μεταρρύθμιση του δικαίου της συμβατικής ιδιοκτησίας η οποία δυστυχώς αντιλαμβάνεστε ότι δεν πέρασε και θέλουμε ακριβώς να έχουν ή δημιουργεί κάποια περισσότερα δικαιώματα απέναντι στις μεγάλες πλατφόρμες. Πώς θέλετε να το προωθήσετε αυτό στο Συμβούλιο για να έχουμε ακριβώς ε, μια ενίσχυση του δημιουργικού τομέα και να βοηθήσουμε και να πληρώνονται οι δημιουργοί στο διαδίκτυο. Εντάξει, κάπως λιγότερο πληρώνονται ήδη για τη μουσική, και ακόμα και αυτό είναι πρόβλημα. Έχουν τελείως διαφορετική διαπραγματευτική θέση οι μεγάλες ε, πλατφόρμες. Ε, έχετε κάποια ιδέα για το πώς μπορούμε να το προχωρήσουμε αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ για αυτήν την ε, ερώτηση. Με απασχολεί εδώ και καιρό, γιατί είμαι πεπισμένος πως ε, το ψηφιακό πλαίσιο μπορεί να αποτελεί πλεονέκτημα για ολόκληρη την ζωή μας, αλλά αρκεί να το χρησιμοποιούμε σωστά. Έχουμε πάρα πολλά επιτεύγματα ε, στην ιστορία της ανθρωπότητας, αλλά ε, δεν τα αντιλαμβανόμαστε απλά ως μία ύπαρξη, αλλά επιβάλλουμε και τους δικούς μας τους κανόνες, κάποιες βασικές αρχές που αναγνωρίστηκαν όπως είπατε σωστά στον αναλογικό κόσμο και πρέπει να εφαρμοστούν ε, και στον ψηφιακό κόσμο. Αν ισχύουν γενικά πρέπει να ισχύουν. Και το θέμα ακριβώς δεν είναι να προστατεύσουμε κάποιο συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο. Θέλω να το πω αυτό Ξεκάθαρα δεν είναι το θέμα να προστατεύσουμε το επιχειρηματικό μοντέλο του τελευταίου αιώνα, αλλά κάποιες βασικές αρχές. Αν κάποιο έχει ιδιοκτησία σε κάτι, αν έχει καταβάλει μια πνευματική προσπάθεια και, και βγάζει λεφτά από αυτό, ε, λογικό είναι ο δημιουργός να λαμβάνει κάτι. Γι' αυτό ακριβώς ε, θα πρέπει και οι μεγάλες πλατφόρμες να επιδείξουν ότι έχουν κάποια προστιθέμενη αξία. Δηλαδή το Google έχει ένα μερίδιο της αγοράς 90% ε, κατ' μιλάμε για ένα μονοπόλιο δηλαδή. Και το τραγικό είναι ότι και οι εθνικές οδηγίες του ανταγωνισμού δεν θα επέτρεπαν, ε, παραδείγματο χάρη, μια ένωση αυστριακών ή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που θα είχαν μια τέτοια ε, συγκέντρωση της αγοράς. Από το 30% και πάνω μιλάμε για δεσπόζουσα θέση. Δηλαδή, εάν προσπαθούσαν να κάνουν ε, κάτι τέτοιο, αυστριακές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν την Google, δεν θα το επέτρεπε η νομοθεσία και το δεχόμαστε για την Google που έχει το 90% της αγοράς. Βλέπετε λοιπόν πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς απευθύνω έκκληση σε όλους ε, στις ε, τριμερείς διαπραγματεύσεις να επικεντρωθούμε σε αυτά. Και όσο το νωρίτερο γίνει τόσο το καλύτερο. Θα πρέπει ακριβώς ε, και τα τρία θεσμικά όργανα να πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Σημαντικό λοιπόν είναι να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Νομίζω ότι σε αυτό το θέμα συμφωνούμε και τα τρία θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέσσερις ομιλητές έχω τώρα και θα κλείσει εδώ πέρα ο κατάλογος γιατί θέλουμε να ακούσουμε και τον κύριο Στράχε, τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως. Σίλβια Κώστα για δύο λεπτά το πολύ. Ναι, για την παρουσίασή σας. Θα μιλήσω Ιταλικά. Ευχαριστούμε, Υπουργέ, που μας παρουσιάσατε και τις προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας και τις προτεραιότητες για τον πολιτισμό. Θα ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια και η Αυστρία στο Συμβούλιο στήριξε το Ευρωπαϊκό Έτος Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς και τα προηγούμενα, τα προηγούμενα χρόνια θελήσαμε να δώσουμε ένα κεντρικότερο ρόλο στην ε, παιδεία, την ε, δημιουργία, την εκπαίδευση στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Γνωρίζετε ότι η νέα ατζέντα για την κουλτούρα, για, την, ε, για τον πολιτισμό, είναι μεγάλη πολιτική προτεραιότητα. Έχουν περάσει 10 χρόνια από την πρώτη τέτοια προσπάθεια, το 2007. Είναι στατηγική ανάγκη να ορίσουμε προτεραιότητες για τα οπτικοακουστικά, τα ψηφιακά, αλλά και για τη δημιουργική Ευρώπη, την Creative Europe, που θα πρέπει να ορίσει, ε, καθότι είμαι εγώ εισηγήτρια και εσείς από την πλευρά της Προεδρίας για τη διπλωματεύση το Συμβούλιο, να ορίσει ε, φιλοδοξότερους στόχους, αλλά ακόμα δεν έχουμε αρκετούς πόρους. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να ξέρουμε αν έχετε σκοπό να επενδύσετε περισσότερο. Κυρίως στο πρόγραμμα πολιτισμός. Μέσα και δημιουργία. 11, 12% μέχρι τώρα δεν είναι αρκετά. Και για, τα, για την ψηφιοποίηση, τα ψηφιακά, όπως είπατε, ισότιμοι κανόνες είναι κάτι το σωστό, αν και η συζήτηση ακόμη στο Κοινοβούλιο δεν έχει ολοκληρωθεί καν, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν αποφάσει για την πνευματική ιδιοκτησία. Είναι απαραίτητη η αναγνώριση των δικαιωμάτων των δημιουργών, αλλά και των, τις αξίες των δημιουργιών που ανατίθενται σε κάποιες επιχειρήσεις. Θα πρέπει η Ευρώπη να προστατεύει όντω, αλλά ο διαπολιτιστικό διάλογο. η στροφή προς την εκπαίδευση και την παιδεία ακόμα και για ανθρώπους που έρχονται από άλλες χώρες νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να ανοίξουμε την Ευρώπη και να μην κοιτάζουμε να την κλείσουμε και να την χειρώσουμε απλώς. Σας ευχαριστώ και εσείς κύριε Μπλίμελ παρακαλώ σύντομα. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε και από τον συνάδελφο. Ναι, ναι, μα μιλάμε τακτικά για την συγκεκριμένη σας ερώτηση για το πρόγραμμα του πολιτισμού και για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το προτινόμενο ύψος. Η Κομισιόν έχει προτείνει κάτι το οποίο θα αποτελέσει οπωσδήποτε την βάση. Υπάρχουν βεβαίως διαφορετικές ε, θέσεις και τα κράτη-μέλη έχουν τις θέσεις τους Ήδη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων είχαμε δύο φορές, δύο γύρους συζητήσεων και εμείς προσπαθούμε ως Προεδρία του Συμβουλίου να έχουμε μια επιτάχυνση των συζητήσεων, όχι μόνο στην Κορεπέρ, αλλά σε κάθε Συμβουλίο Γενικών Υποθέσεων συζητιέται το θέμα αυτό γιατί ακριβώς υπάρχουν κάποιες προσδοκίες ότι ίσως θα καταλήξουμε σε κάποια απόφαση πριν από τις ευρωεκλογέ. Αν δείτε τις τελευταίες συζητήσεις, βεβαίως ε, τις τελευταίες φορές, πάντα διαρκούσε λίγο περισσότερο αυτή η διαδικασία, αλλά έχουμε κάποια φιλοδοξία. Τώρα, είναι διαφορετικές οι εθνικές θέσεις ε, και η κατάσταση της ε, συζήτησης ε, και η πρόταση της Κομισιόν είναι μια πρόταση αρκετά θετική, αλλά τώρα δεν μπορώ να προδικάσω το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ χιλικά Τρίπελ. Ευχαριστώ Πέτρα να αναφερθώ στη μεταρρύθμιση του δικαίου της ε, πνευματικής ε, ιδιοκτησίας. Δεν πρέπει μόνο να δούμε κάποιο νέο business model, αλλά να υπάρχει η δυνατότητα να έχει κάποιος ε, business model, γιατί υπάρχουν τα lobby της Google και λοιπόν που λένε ότι υπάρχει μια γενική λογοκρισία και ένας φόρος ε, στα link. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν, τα ιδιωτικά link ε, δεν ε, έχουν καμία τέτοια αντιμετώπιση. Θέλω λοιπόν να είναι ξεκάθαρο. Είναι λοιπόν απολύτως απαραίτητο γιατί ακριβώς έχουμε από τη μία τις μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις και από την άλλη τους καλλιτέχνες και πρέπει να προστατεύσουμε τους μικρούς από τους μεγάλους. Γι' αυτό ακριβώς κάνουμε πολιτική. Κύριε Υπουργέ, όχι. Το να ακούω εδώ πέρα εκκλήσεις ε, είναι θετικό. Αν διαβάζατε το πρόγραμμά μας ε, θα βλέπατε ότι ακριβώς θέλουμε ε, να δίκαιο προστασίας των δημιουργών. Ιδανικά λέμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εάν δεν γίνει αυτό σε εθνικό επίπεδο, γιατί θεωρούμε ότι η ιδιοκτησία πρέπει να προστατεύεται ψηφιακή ή αναλογική. Ελπίζω λοιπόν να καταλήξουμε σε μια συζήτηση το στομότερο δυνατόν ε, στο Κοινοβούλιο γιατί ακριβώς αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί, ότι θέλουμε δηλαδή δίκαιες συνθήκες στην ψηφιακή σφαίρα όπως και στον αναλογικό χώρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ είμαι Τσέχα. Δύο μόλις ώρες από τη Βιέννη, στη Μοραβία. Και όντω οι πολιτιστικέ μα ρίζε και προτάσει είναι ο πλούτο τη Ευρώπη. Νομίζω ότι και γι' αυτό ακριβώ το λόγο η Δημοκρατία τη Τσεχία ξεπέρασε την περίοδο του κομμουνισμού. ένα απόσπαστο τμήμα τη Ευρώπη. Αυτή η πολιτιστική λοιπόν ποικιλομορφία μα βοηθάει. Και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει να μα βοηθάει και στο μέλλον. Ε, Σταθήκατε σε ένα σημαντικό σημείο, μια δραστηριότητα σημαντική του Ευρωκοινοβουλίου και ήθελα και εγώ να το τονίσω. Το βραβείο Lux για τον κινηματογράφο. Το βραβείο Lux είναι σημαντικό διότι η Ευρώπη θα πρέπει να στραφεί και στους Ευρωπαίους ε, δημιουργούς. Θέλουμε να βραβεύσουμε ε, ταινίες, φιλμ που εκτιμώνται, όχι μόνο εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, μάλιστα πολύ συχνά οι βραβευθέντες είναι και από την Αυστρία. Να φροντίσουμε λοιπόν να γίνει πιο γνωστό αυτό το βραβείο μαζί με τις ταινίες που συμμετέχουν. Μιλάμε για ταινίε που έχουν πολλές φορές και υποτιτλισμό, οπότε μπορούν να τις δουν όλοι οι πολίτες και αυτό θα μπορούσε να ενταχθεί στι δραστηριότητε τη ε, Δημιουργική Ευρώπη. Τα φεστιβάλ, τα κινηματογραφικά φεστιβάλ είναι καλό να ε, υποστηρίζονται ώστε τα ε, ταινίε να έχουν την απαραίτητη στήριξη. Το Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι για το ότι είμαστε γείτονες. Έχω και ρίζες από την Τσεχία, η γιαγιά μου ήταν από την Σουδητία και μετά την πτώση του παραπετάσματος ξαναπήγαμε στην ε, γενέτειρά μας ε, και καλό είναι ακριβώς ε, το να περνάμε τα σύνορα και να το δούμε αυτό το θέμα των εσωτερικών σύνορων της Ευρώπης. Λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερος για το ότι η οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα έχει κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός και για το ότι στις μεγάλες πλατφόρμες θα πρέπει πλέον να υπάρχει και ευρωπαϊκό περιεχόμενο έως και 30% Λοιπόν, Ακριβώς ε, βλέπουμε το τι γίνεται και στην ε, Αυστρία με το Netflix που δείχνει αυτή τη σειρά για τους μεδίκους ε, πάρα πολύ συναρπαστική για την ευρωπαϊκή ιστορία και ένα εξαιρετικό παράδειγμα και νομίζω ότι χρειαζόμαστε και άλλα τέτοια και θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε και άλλα τέτοια μέσω των προτάσεων μας στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. και κυρία Κάπελ σύντομα. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ενθαρρύνω εκεί όπου σταμάτησαν ακριβώς οι δύο συνάδελφοι το θέμα του copyright είδαν πόσο σημαντικό είναι. γιατί αναπέμφθηκε η πρόταση τελικά και δεν πήγε στον τριμερή διάλογο. Γι' αυτό ακριβώς ε, θα πρέπει να μην τα αφήσουμε αυτά μόνο στους ε, μεγάλους γίγαντες ε, του διαδικτύου. Είχαμε εδώ πέρα και τον Επίτροπο ο οποίος μας είπε ότι θα πρέπει ακριβώς να δούμε ποια είναι τα περαιτέρω βήματα και ίσως θα μπορούσε και η Κομψιό να κάνει κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν και η Κομισιόν να βρει μία προσέγγιση για να έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά αυτό το κενό της αξίας. Δεύτερο θέμα, το Creative Europe, το πρόγραμμα αυτό πρόθεσης ε, του δημιουργικού κλάδου. Θεωρώ ότι κάτι το οποίο ήταν ε, σημαντικό και θα πρέπει να δικτυωθεί και με άλλα προγράμματα, με τα διαρθρωτικά ταμεία και του ορίζοντα 2020. Νομίζω ότι μας βοηθάει για την δημιουργία προσθέμενης αξίας. Ε, τρίτο, για την πολιτική κληρονομιά, πράγματα τα οποία επίσης ως ε, δέσμες ε, και ως κόμβι είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τον τουρισμό, το ουσιαστικό εδώ πέρα κάτι το πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι ένα πλεονέκτημα που έχει η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ και εσείς σύντομα παρακαλώ, κύριε Μπλούμελ. Για το θέμα του copyright το είπα πολλές φορές. Βεβαίως. Η πολιτική κληρονομιά είναι σημαντική και για τον πολιτισμό και για την χώρα μας και το θέμα είναι ακριβώς πώς θα την προωθήσουμε και να έχουμε μια στρατηγική όχι μόνο για την προστασία της αλλά να αναπτυχθεί μια προστιθέμενη αξία. Και βεβαίως έχουμε την διάσκεψη του πολιτισμού για την Ευρώπη που θα έχουμε στην Βιέννη τον Δεκέμβριο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε λοιπόν με αυτό το κομμάτι της συνεδρίασής μας. Ευχαριστούμε κύριε Μπλούμελ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, και για την κατανόηση. Περνάμε τώρα στον κύριο Στράχε. Έχετε λοιπόν αμέσως τον λόγο για τον τομέα του αθλητισμού. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε κυρίες και κύριοι βουλευτές. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να αναφέρω τις προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας στον τομέα του αθλητισμού. Θα μας απασχολήσουν λοιπόν τα εξής θέματα. Ουσιαστικά η οικονομική διάσταση του αθλητισμού και εδώ πέρα βεβαίως ε, θα αναδείξουμε την οικονομική σημασία του αθλητισμού, το πώς συνεισφέρει στην οικονομία της Ευρώπης και πώς μπορεί ακριβώς να βοηθήσει την ανάπτυξη, την απασχόληση και ταυτόχρονα βεβαίως ο αθλητισμός είναι και μία εγγύηση και για την γενικότερη ευημερία των λαών μας. Ε, το μετρήσει κανείς, μιλάμε για ένα 2% του ΑΕΠ, στην Αυστρία είναι ένα 7% μάλιστα. Αυτό δείχνει ακριβώς την διάσταση που μπορεί να δημιουργηθεί σε περιφερειακό επίπεδο. Ε, το σημαντικότερο κομμάτι δε στην Αυστρία είναι ο τομέας ε, των οικοδομών για να πάρετε μια εικόνα. Και βεβαίως Έχουμε και τους Ολυμπιακούς προσεχώς το 2024 στο Παρίσι. Οπότε έχουμε μια σημαντική ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας στη δε Αυστρία του χρόνου θα προετοιμάσουμε ε, ακριβώς ε, ένα τεχνικό ίδρυμα για τα χειμερινά σπορ. Βεβαίω το θέμα αυτό είναι κάτι το οποίο αγγίζει τα πάντα. Την υγεία, την πρόληψη, τα μικρά παιδιά, την οικονομία και τον τουρισμό. Η οικονομική διάσταση, όπως σας είπα, σχετίζεται με την έρευνα και την ε, καινοτομία. Στόχος λοιπόν είναι να υιοθετηθούν αυτά τα συμπεράσματα από το Συμβούλιο του Νοεμβρίου. Κάτι άλλο σημαντικό, όπως είπα, θα είναι ο αθλητισμός και η υγεία. Η Αυστριακή Προεδρία θα ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, θα δώσει ιδιαίτερο βάρος ε, στην υγιεινή, στην εργασία και θα οργανώσουμε και ένα σεμινάριο ειδικών στις 10 Δεκεμβρίου στην Βιέννη όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές, να ανταλλάξουμε εμπειρίες, να δούμε το τι μπορεί να γίνει στο χώρο εργασίας, σκάλες αντί για σανσέρ κτλ. Και επιπλέον βεβαίως έχουμε τον αγώνα καταπολέμησης του ντόπινγκ που είναι ένα θέμα που είναι διαρκώς ε, σημαντικό. Είχαμε τα τελευταία σκάνδαλα με τους Ρώσους κυρίως αθλητές που δημιουργήσαν πολύ αρνητικούς ε, τίτλους. Ε, άρα είναι κάτι το πολύ σημαντικό και ακριβώς τώρα έχουμε την δεύτερη φάση ε, της, δεύτε, της παγκόσμιας διάσκεψης κατά του ντόμπινγκ και βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό Αυστριακή Προεδρία θα συνυπογράψει αυτές τις ε, προδιαγραφές. Επίσης θα δούμε και το μέλλον του παγκοσμίου συστήματος καταπολέμησης του ντόπινγκ και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παρακολουθεί αυτήν την συζήτηση από κοντά και οπωσδήποτε αυτά θα δούμε και με τη Γουάντα, την ε, Παγκόσμια Υπηρεσία Καταπολέμησης ε, του Ντόπινγκ. Επιπλέον ε, έχουμε και τον συντονισμό με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Γουάντα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το πρόγραμμα Erasmus Plus ένα από τα πιο επιτυχή προγράμματα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα αυτό της κινητικότητας είναι από τα πιο αγαπητά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα ένα σύμβολο για την Ευρώπη και τις αξίες μας. Το 2014 λοιπόν έχουμε το αθλητικό τμήμα του προγράμματος που ξεκίνησε την εισαγωγή μικρών συνεργασιών ε, και το 2016 είχαμε αύξηση του αριθμού των προγραμμάτων και η Κομισιόν οπωσδήποτε θα υποβάλει την πρότασή της για το μελλοντικό πρόγραμμα Erasmus Plus, κινητικότητα προπονητών ε, και αθλητών. Ε, θα παίξει έναν βασικό ρόλο το θέμα λοιπόν είναι ακριβώς η κινητικότητα της εκπαίδευσης των μαθητών και αυτό το οποίο είπε και ο συνάδελφος να υπάρχει η μετάβαση και στον χώρο εργασίας. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τις προτάσεις μας και είμαστε σίγουροι ότι θα επιτύχουμε κάποιες ε, συμβιβασμούς και κάποια αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν και την διάσκεψη των ειδικών ε, που θα συγκαλέσουμε με θέμα την οικονομική διάσταση του αθλητισμού, την συνεισφορά της στην απασχόληση. 21 Σεπτεμβρίου 2016 θα γίνει με την άτυπη συνάντηση των διευθυντών αθλητισμού. Ο αθλητισμός ε, και η σωματική άσκηση θα αποτελέσει θέμα ε, επίσης σεμιναρίου στη Βιέννη και θα έχουμε και τη μεγάλη εβδομάδα αθλητισμού 26 ε, Σεπτεμβρίου που βεβαίως θα χαρώ να σας δω και εσάς ε, στην Βιέννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αντιπρόεδρε της κυβερνήσεως. Λοιπόν, έχουμε τον Μπόγκταν εδώ, τον ιδρικό του αθλητισμού. Ε, σε παρακαλώ όμως να έχεις κατά νου και το χρόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω λοιπόν να τα πω κι εγώ στα γερμανικά. Αξιότιμε, κύριε Αντικαγκελάρια, χαίρομαι για τις προτεραιότητες που μας αναφέρατε, για το όραμα, για την οικονομία, στον αθλητισμό. Ε, μιλήσατε και για την υγεία. Προφανώς είναι σημαντικό. Το ντόπινγκ επίσης. Κι εγώ είμαι πρώην αθλητής και είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε το, τη μάστιγα αυτή. Το Erasmus Plus Ούτως ή άλλως είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει και σήμερα και γενικώ μας απασχολεί όλους. Το ερώτημά μου είναι σύντομο και απλό. Για αυτές τις τέσσερις προτεραιότητες που μας αναφέρατε. Είπατε κάτι για τις διασκέψεις και τις διάφορες ημερίδες, αλλά κάποια συγκεκριμένα μέτρα κατά τη διάρκεια της α, Προεδρία προτίθεστε να πάρετε και μετά επειδή είμαι και ο εισηγητής για τη χειραγώγηση στον αθλητισμό, υπάρχει και η, ε, ειδική σύμβαση από το Συμβούλιο της Ευρώπης και εκεί Υπάρχουν αρκετά ευρωπαϊκά κράτη που ε, υποστηρίζουν την πρωτοβουλία αυτή, πολλά εκ των οποίων είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχει και ένα αδιέξοδο. Μία χώρα μπλοκάρει την όλη διαδικασία, η Μάλτα συγκεκριμένα. Και το ερώτημα είναι απλό. Νομίζω ότι μπορούμε από κοινού κάτι να κάνουμε, γιατί θα ήταν καλό το μήνυμα προς τα έξω. αλλά η δική σας άποψη ποια είναι για το θέμα αυτό και η Αυστριακή Προεδρία τι μπορεί να κάνει σε αυτόν τον τομέα. Γιατί εγώ ως συζητητής δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είμαι μπλοκαρισμένος αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Αντικαγκελάρια. Αξιότιμη κύριε Βέντα. Ευχαριστώ για τις διαπιστώσεις και για το ερώτημά σας. Ο αθλητισμός είναι ένας τομέας που περιλαμβάνει πολλά και προσπαθούμε να φέρουμε τον αθλητισμό πιο κοντά στους πολίτες, να τους ε, εξοικειώσουμε με την κίνηση, με την άσκηση προσπαθούμε όλα αυτά να τα δημιουργήσουμε και εντό τη ε, δική μα χώρα και βεβαίω υπάρχει μεγάλη σημασία και να γίνει αυτό και μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και για τον απλό πολίτη που μπορεί να μπει στον, στον, τομέα του αθλητισμού, αλλά και για τους πρωταθλητές και για τους επαγγελματίες αθλητές. Τώρα, για τη χειραγώγηση στα, στα σπορ και το match fixing, υπάρχουν ε, όντως πολλοί τομείς, ε, πολλά είδη αθλητισμού που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδου σκάνδαλα. Και το τελευταίο, στο τελευταίο σκάνδαλο δυστυχώς ε, πλήγει το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό ισχύει και για άλλους τομείς. Εμεί ε, παρακολουθούμε τις διεθνεί εξελίξεις πολύ προσεκτικά και δείχνουμε μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως ε, για την σύμβαση κατά της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων των, του αθλητισμού και ε, είχαμε υποβάλει την συγκεκριμένη συμφωνία για το 2015 τώρα και το 2017 υπάρχουν προτάσεις ακριβώς για την υπογραφή της, ε, την ολοκλήρωση ας πούμε της σύμβασης αυτή η Προεδρία θα εξετάσει πώς μπορούν να, προωθήσουν, να προχωρήσουν αυτές οι προτάσεις στο Συμβούλιο Βεβαίω είναι σημαντικό να το πετύχουμε αυτό, κυρίω για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτή την σύμβαση. Αλλά βεβαίω πρέπει να είμαστε και ε, ρεαλιστέ. Στο παρελθόν δεν μπορέσαμε να έχουμε συμφωνία για τη σύμβαση αυτή. Αν δούμε τώρα και την ε, κατάσταση στο Συμβούλιο, ε, ίσω να είναι λίγο δύσκολο να επιφέρουμε πρόοδο. Οπότε είμαστε κι εμεί λίγο, λίγο με δεμένα τα χέρια. Θα παρακολουθούμε βέβαια την κατάσταση και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια κοινή λύση. Και μετά ε, για τις εκδηλώσεις ε, που είπατε, 22 Σεπτεμβρίου 2018, η Εθνική ημέρα του αθλητισμού στην Αυστρία. Και εκεί θα εισαχθεί, μάλλον θα ξεκινήσει και η εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Ευχαριστώ ίσως ε, να καταφέρετε εσείς με τη Μάλτα αυτό που δεν κατάφεραν οι προηγούμενες ε, προεδρίες. Ίσως να καταφέρετε να πείσετε εσείς να μετακινηθεί λιγάκι η Μαλτέζια κυβέρνηση. Χέλικα να ρωτήσω κάτι για, το, για την αντιμετώπιση του ντόπινγκ. Εγώ είμαι 14 χρόνια εδώ και κάθε φορά το συζητάμε ότι και λέμε ότι πρέπει να κάνουμε κι άλλα. Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, πρέπει να γίνουμε ε, πιο επαρκείς. Και Θέλω να ρωτήσω, εσείς έχετε συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί έχουμε την ε, ε, ιστορία ε, αυτού του δημοσιογράφου στη Ρωσία που αποκάλυψε το σκάνδαλο και μετά αναγκάστηκε να εξαφανιστεί γιατί δεν λάμβανε απειλές για τη ζωή του. Έχετε εσείς λοιπόν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για το τι μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της δικής σας προεδρίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε, εκπροσωπούνται σε επίπεδο υπουργών, όπου λαμβάνονται συνήθως τα μέτρα. Υπάρχει και η εκπροσώπηση στο, στην Τρόικα των Προεδριών. Μέχρι στιγμή ο Υπουργός της Βουλγαρίας, ο Υπουργός Αθλητισμού, είναι σε, είμαστε, είναι σε επαφή μαζί μας και με, εμείς είμαστε και σε επαφή με τον Υπουργό της Ρουμανίας, Υπουργό Αθλητισμού. Αυτοί εκπροσωπούν την ευρωπαϊκή μας ε, θέση και στην Γουάντα. Και βεβαίως φυσικά θέλουμε και εμείς εδώ να έχουμε κοινού κανόνες, οι οποίοι βεβαίως να είναι σε συνάφεια και με τους ε, διεθνείς κανόνες και βεβαίως θα το παρακολουθούμε, αλλά βεβαίως πρέπει να δούμε εκεί που γίνονται παραβάσεις και παραβιάσεις ε, να υπάρχουν και απαραίτητε συνέπειες. Κυρίως για τον τομέα του ντόπινγκ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπίλτ. Παρακαλώ, ναι. έχετε υπόψη σας και το χρόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για την ε, προσέλευσή σας σήμερα το πρωί και συγχαρητήρια για τις πρώτες ε, κατευθύνσεις που μας έχετε διαγράψει, περιγράψει. Ε, για ένα θέμα που μας απασχολεί το 2017-2018, το Erasmus συν Ασκή και δράσεις, υλοποιεί και ασκήσεις, δράσεις ένταξης κυρίως για πρόσφυγες και μετανάστες. Με το πρόγραμμα Κόρπλε, ας πούμε, γιατί μέσω του αθλητισμού σκοπεύουμε να ενσωματώσουμε και τους ε, αλλοδαπούς. Σας φαίνεται ότι αυτό συνάδει με το πνεύμα του Εράσμου Συν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Βουλευτά. Ε, το Erasmus Plus, εντάξει, ό,τι έχει να κάνει με τον ε, αθλητισμό, ένωση των λαών, ένταξη, συμμετοχή. Νομίζω ότι χρειάζεται το δικό, της, το δικό του πρόγραμμα α, χρηματοδότησης. Ο αθλητισμός ε, ούτως ή άλλως είναι μια θετική ανταλλαγή και συμμετοχή, με συμμετοχή όλων από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αν τώρα μιλούμε για την ε, συμμετοχή, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό η ένταξη, η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στον αθλητισμό. Και εκεί θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε πιο εντατικά για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουν και αυτοί, θα μπορούν να υποφεληθούν από την ισότητα αυτή. Να μπορούν να συμμετέχουν όπως όλοι οι υπόλοιποι αθλητές. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε στον πυρήνα των συζητήσεών μας, ε, γιατί ούτως ή άλλως και το Erasmus Plus είναι ένα πρόγραμμα ένταξης. Περιλαμβάνει δηλαδή αυτή την ε, σύγκληση. Ευχαριστώ. Δύο ακόμα παρεμβάσεις έχω. Δεν μπορώ να σας ε, δώσω και το, το λόγο και στους δύο, γιατί και οι διερμηνείς ε, βρίσκονται σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορούν να μας δώσουν περισσότερο χρόνο. Οπότε, να, δεν μπορώ να δώσω το λόγο σε άλλους πια. Σας ευχαριστώ. Κυρία Αντικαγκελάρια Στράχη, κυρία Υπουργέ Μπλούμελ, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ σήμερα. Νομίζω είδατε κι εσείς ότι είμαστε μια πολύ αφοσιωμένη στα θέματά μας επιτροπή. Κυρίως όταν μιλούμε για θέματα οικονομικά βεβαίως ε, ε, δεν είναι και πολύ διασκεδαστικά τα θέματα, αλλά δεν είναι όσο διασκεδαστικό είναι ο αθλητισμός και η νεολαία. Ελπίζω ότι θα έχουμε στο πλευρό μα την Αυστριακή Προεδρία για τα θέματα αυτά και βεβαίω σας εύχομαι κάθε επιτυχία για, την, για το επόμενο εξάμεινο της Προεδρία. σας. Ευχαριστώ.